Κυρίε Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner votre place, s'il vous και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Θα ήθελα καταρχάς να σας καλωσορίσω σε αυτήν την ε, Διακοινοβουλευτική Επιτροπή και να σας ευχαριστήσω που ε, επιλέξατε αυτή την συνεδρία της οποίας ηγείται η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου και εγώ ως πρόεδρος αυτής της Επιτροπής έχω το προνόμιο να ξεκινήσω αυτή τη συνεδρίαση τη διακοινοβουλευτική. Οι σχέσεις μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντείνονται και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να έχουμε μια ειδική σχέση με την Επιτροπή που ασχολείται με τα οικονομικά και με τον προπολογισμό συγκεκριμένα στα Εθνικά Κοινοβούλια. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου. Σήμερα το πρωί στην Ολομέλεια, η Ολομέλεια υπόθηκε ότι δεν πρέπει να υπερεκτιμούμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό είναι το 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Αυτός ο προϋπολογισμός είναι, περιβάλλεται από ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 7 ετών, το οποίο ξεκίνησε το 2014 και θα ολοκληρωθεί το 2020. Οι πόροι για, τα βασικά, για τις βασικές δαπάνες προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Οπότε ο καθένας πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη για να δώσει τον οβολό του για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ήδη πόρη είναι 10% και όπως είπε ο Μάριο Μόντι θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο το θέμα των ίδιων πόρων σε θεσμικό επίπεδο δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα αν μπορούσε να ψηφίσει ε, για τη φορολογία κάτι που στην ουσία θα ήταν θεσμική Θα Θεωρούμε λοιπόν ότι θα ήταν ένας ε, φόρος ευρωπαϊκός ο οποίος ε, θα προστίθετο στους εθνικούς φόρους και αν υπήρχε ένας τέτοιος φόρος δεν θα έπρεπε να επιβαρύνει επιπλέον τους Ευρωπαίους φορολογούμενους έτσι ώστε να μειωθούν οι εθνικές φορολογίες. Αυτό το πλαίσιο λοιπόν στην ουσία μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε πόρους στα κράτη-μέλη μέσα από πιστώσεις ε, ε, σύγκλησης και το 80% των πιστώσεων πραγματικά πηγαίνουν προς τα κράτη-μέλη στην ουσία δεν υπάρχει περιθώριο ευελιξίας. Ε, έπρεπε αυτό να χρησιμοποιηθεί σε νηνεμία. Όμως τώρα έχουμε μια εξαιρετική κατάσταση και οι Ευρωπαίοι αναρωτιούνται τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολύ περιορισμένοι πόροι. Όταν ήρθε ο Γιούνκερ στην Προεδρία της Κομισιόν διαπίστωσε κάτι πολύ Σημεριζόμαστε ότι εδώ και 10 χρόνια η Ευρώπη έχει ένα έλλειμμα επενδύσεων και πρέπει να ενισχύσουμε τις επενδύσεις. Και υπήρξε ε, ένας μηχανισμός ε, μόχλευσης ε, που στην ουσία επινοήθηκε για να μπορέσουμε να έχουμε στρατηγικές επενδύσεις, να δώσουμε δηλαδή χρήματα έτσι ώστε να υπάρχουν εγγυήσεις για κονδύλια. Και δυστυχώς στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου έπρεπε να δούμε ότι στον ορίζοντα 2020 και το ε, Connecting Europe Facility που είναι υπερεθνικές επενδύσεις έπρεπε να γίνουν περικοπές. Όμως για να βρούμε μερικές ε, δεκάρες δεν έπρεπε να πάρουμε χρήματα από τα κράτη-μέλη, έπρεπε να πάρουμε από τους πόρους που είναι υπερεθνικοί για να μην έχουμε τους ε, εθνικούς εγωισμούς. Έτσι λοιπόν το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο εγκρίθηκε πριν την ανανέωση της θητείας του Κοινοβουλίου. Ήταν δηλαδή στη θητεία του 2014 και βλέπετε ότι κάθε χρόνο ο προπολογισμό είναι ένα κομμάτι αυτού του πλαισίου, του δημοσιονομικού. Στις συζητήσεις τότε υπόθηκε ότι και συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί αυτό το πλαίσιο ε, στη μέση του, να λάβουμε υπόψη τις περιστάσεις, γιατί είναι λίγο αναχρονιστικός ο προϋπολογισμός που έχουμε τώρα. Δεν μας δίνει τα μέσα να αντιμετωπίσουμε τα νέα στοιχεία. Αυτό που διαπιστώθηκε και με τις επενδύσεις. Έπρεπε να δημιουργηθεί ένα ειδικό εργαλείο εκτός του προϋπολογισμού που θα πιλωτάρεται, ας πούμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από εκεί θα καθοδηγείτε. Ε, τώρα που έχουμε την μεταναστευτική κρίση και τους πρόσφυγες ε, έχουμε νέες ανακοινώσεις για ένα trust fund που θα έχει πιστώσεις πάλι από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και από τη Γενοδορία των Κρατών Μελών στην οποία κάναμε έκκληση. Οι μεταφορές αυτές πόρων ε, ε, θα γίνουν βάσει του πλαισίου που έχουμε το 2014 και όσον αφορά την Τουρκία και τις ανακοινώσεις που έγιναν ε, για τα ε, δις που ανακοινώθηκαν για το Φλεβάρι του 2016 υπήρχαν 40 εκατομμύρια. Έτσι λοιπόν ανακοινώθηκαν τρία δις για την Τουρκία για να μπορεί να υποστηρίξει τους ε, πρόσφυγες που έρχονται σε μεγάλους αριθμούς από τη Συρία. Οπότε πρέπει να βρεθούν τα μέσα για να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση αυτής της υπόσχεσης. Τώρα στην ε, προπαρασκευαστική φάση της αναθεώρησης του ε, του δημοσιονομικού πλαισίου βάζουμε και τη βάση για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και πρέπει να δούμε αν αυτό το 7 ετές πλαίσιο θα μπορέσει να γίνει 5 Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή την αναθεώρηση, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, ε, έχει δύο ε, οι εισηγητές, την κυρία Τομά από τους Σοσιαλιστές και τον κύριο Ολμπρί από το ΕΛΚ, ο οποίος σήμερα δυστυχώ δεν είναι εδώ. Οπότε η κυρία Ιζαμπέλ Τομά από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες ε, θα μας μιλήσει για τις προπαρασκευαστικέ εργασίες αυτής της αναθεώρησης του ΠΙΒΕΛΤΑΠΗ για να μπορούμε να έχουμε ένα σχέδιο ψηφίσματος πριν το τέλος του 2016 που θα γίνει η τελική αναθεώρηση για να δούμε αν θα υπάρχουν περισσότεροι, περισσότεροι πόροι, περισσότερες πιστώσεις. Κάτι που δεν το βλέπουμε και αν δεν υπάρχουν και υπάρχουν έκτακτες ανάγκες θα πρέπει να γίνουν πολύ σημαντικές μοχλεύσεις και αναδιαπραγματεύσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το σχέδιο του 2014-2020. Έχουμε λοιπόν την πρώτη ώρα αφιερώσει σε αυτό το θέμα. Θα γίνει μια συζήτηση και αυτοί που θα λάβουν το λόγο ζητώ να μιλήσουν μέχρι και δύο λεπτά για να μπορέσουμε να μιλήσουμε όλοι. Στις τέσσερις θα γίνει πάλι μια δεύτερη συνεδρία. Θα δούμε ε, Ποιε θα είναι οι προτεραιότητες για το ΠΔΠ 2014-2020 και τις νέες ε, οικονομικές ανάγκες για την κρίση των προσφύγων. Μία ώρα θα αφιερώσουμε σε αυτό το θέμα και άλλη μία ε, ώρα έχουμε για τις οικονομικές ανάγκες που χρησιμοποιούνται για να ξεπεράσουμε την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση. Έχουμε το παράδειγμα Τη πρωτοβουλία ε, για την απασχόληση των νέων. Η κυρία Τομά έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ που είστε παρόντες όλους. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει καθ' όλη τη διάρκεια του 2016, γιατί όπως είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, Προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε νομικό πλαίσιο τα πράγματα είναι απλά αλλά σε πολιτικό επίπεδο δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Σε νομικό επίπεδο ξέρετε ότι ψηφίζουμε ετησίως τον προπολογισμό, αλλά σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο που είναι πολιετές, που εδώ και πολλές δημοσιονομικές χρήσεις διαρκεί 7 χρόνια. Φαντάζεστε τι μπορεί να συμβεί μέσα σε 7 χρόνια. Σε νομικό επίπεδο λοιπόν έχουμε αυτό το δελτα για 7 χρόνια ε, για αυτή την περίπτωση έχουμε, ξεκινάει το 2014 μέχρι το 2020 με τους α, κλειστούς φακέλους για τη συνοχή, δηλαδή δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε αυτά, με ένα, μια ανώτατη οροφή για τις ε, δαπάνες πολύ συγκεκριμένη που σαν ήδη και κάποια στοιχεία έτσι λίγο ξεχαρβαλωμένα ευελιξίας και κάποιες λειτουργίε στις οποίες θα επανέλθουμε. Στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013 το Κοινοβούλιο είχε διαπιστώσει την ανάγκη για μια τόσο μακροσκελή περίοδο να αναθεωρηθούν οι οροφές, η ευελιξία του προϋπολογισμού, κάτι που δεν προβλεπόταν ε, επαρκώς και ακριβώς γι' αυτό όταν θελήσαμε να ψηφίσουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο 14-20, εμείς είχαμε βάλει κάποιες προϋποθέσεις ως Κοινοβούλιο, μεταξύ των οποίων το άρθρο 2, το οποίο προέβλεπε ότι μπορούμε να αναθεωρήσουμε ή να επανεξετάσουμε το πλαίσιο αυτό στα μέσα της διαδρομής, στα μέσα της πορείας. Και πιο συγκεκριμένα έλεγε πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2016, πριν το τέλος το φετινό δηλαδή, Τη φετινή χρονιά, η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει πρόταση. Ε, μια και είχαμε καεί στο χυλό, φορούσα, ε, φοβόμασταν ότι η Κομισιόν θα καθυστερήσει και η Επιτροπή Προπολογισμών μέσω του Προέδρου πρότεινε να γίνει μια έκθεση πρωτοβουλία για να προετοιμάσει τη θέση του Κοινοβουλίου. Φυσικά, τώρα το θέμα, όπω είπε και ο πρόεδρο είναι πού έχουμε φτάσει. Όχι πολύ μακριά. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε φυσικά τι θα ψηφίσει το Κοινοβούλιο μετά τις συζητήσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει μάλιστα, και την ψηφοφορία που θα γίνει το πρώτο εξάμεινο του 2016, κατά πάσα πιθανότητα τον Ιούλιο. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα απ' την άλλη, το υπενήθηκε και ο Πρόεδρος, το πλαίσιο είναι πλαίσιο πολλαπλών κρίσεων, πολύ περισσότερο από την προηγούμενη χρονιά, την προηγούμενη περίοδο προϋπολογισμού, είμαστε στο χείλος της Αβίσου, να το πούμε αυτό. Ε, και αισθανόμαστε μια μεγάλη αδυναμία, όχι ολική, για την κρίση ας πούμε την, ε, των προσφύγων, ε, έκρηξη του Σέγγεν, ε, απειλούμαστε από πολλαπλές διαιρέσεις, α, αποχωρήσεις ε, κατών μελών. Χθε είχαμε τον Brexit, χθες προχθές είχαμε τον Brexit, τώρα αύριο μεθαύριο έχουμε το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω λοιπόν, θα πρέπει να προσθέσω τις λεγόμενες επαναλαμβανόμενες κρίσεις προϋπολογισμού τη Ένωση, διορθώνει ομιλήτρια. Δηλαδή ψηλό επίπεδο ανεργία, δραματικό στους νέου, 25% των νέων κάτω των 25 χρονών είναι άνεργοι. Άλλη επαναλαμβανόμενη κρίση, το είπε και ο πρόεδρο, είναι το θέμα των επενδύσεων. Πολύ χαμηλέ επενδύσει. Η χρηματοπιστωτική κρίση με νέε απειλέ σήμερα και κάτι που δεν ξέρω τόσο καλά είναι η κρίση των πληρωμών είναι μια ειδικότητα του προπολογισμού της Ένωσης αυτή, η οποία ε, δεν πρέπει να είναι ελληματική, όπως το, ο προπολογισμό δηλαδή όπως ξέρετε, δεν έχουμε δικαίωμα, το λέει η συνθήκη, αλλά έχουμε ε, πολύ πιο ψηλές δεσμεύσεις από πληρωμές. Ε, και το Δεκέμβριο του 2014 φτάσαμε όχι σε χρέωση, αλλά είχαμε 24 δις ε, λογαριασμών απλήρωτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς να το πω. Χρέωση, έλλειψη πληρωμών. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να φτάσουν στους προπολογισμού των ε, τοπικών αρχών, ε, στις ε, επιχειρήσεις, στα, στους φοιτητές του έρασμου, στα εργαστήρια κτλ. Κάπου στους δικαιούχους τέλο πάντων. Αυτά τα 24 δις. Αυτή είναι, αυτό είναι το πλαίσιο της κρίσης που είναι και διαφθορτικό και συγκυριακό ε, και θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Δυστυχώς αυτές οι αποφάσεις πρέπει να το ομολογήσουμε. Δεν έχουν ληφθεί στην πραγματικότητα. Δεν πιάσαμε τον τάβρο τα κέρατα και θα πρέπει να προσθέσουμε ότι μία από τις αιτίες, όπως είπε και ο Πρόεδρος, είναι ότι το 80% περίπου του προπολογισμού της Ένωσης αποτελείται από επιταγές των κρατών μελών και κατά συνέπεια ε, το κλασικό ανακλαστικό που έχουν όλοι οι εθνικοί βουλευτές και εδώ θα γίνει συζήτηση, και οι κυβερνήσεις είναι να περιορίσουν όσο πιο χαμηλά γίνεται να συμπιέσουν αυτή την εκροή για να κρατήσουμε μεγάλο περιθώριο ελιγμού στον εθνικό προπολογισμό. Το καταλαβαίνουν αυτό. Δεν είναι κατηγορία. Ούτε εδώ ας πούμε αδεικνύουμε τους εγωισμούς. Απλώς είναι μια δομή ας πούμε δημοσιονομική που οδηγεί σε τέτοια ανακλαστικά. Παρ' όλα αυτά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε μία μορφή δημοσιονομικής ανηλικρίνειας, για να το πω έτσι. Γιατί τα κράτη-μέλη, και εδώ θα περάσω σε πιο άμεση, ας πούμε, σε πιο άμεσο κατηγορό. Τα κράτη-μέλη, μόλις εμφανίζεται μια κρίση, δεν διστάζουν να πούν «Α, εδώ θα βάλουμε τέσσερα δίστη για την Τουρκία, τρία δις, ας πούμε, από την άλλη για την υποδοχή των προσφύγων, 8 δις ε, για το Ταμείο Επενδύσεων του σχεδίου Juncker, κουλουπού κουλουπού. Δηλαδή, από, την από τη μία δεν βάζουμε λεφτά στο κουμπαρά και μάλιστα βάζουμε όσο το δυνατόν πιο λίγα και από την άλλη δεν διστάζουμε όταν υπάρχει μια δεν βαζουμε λεφτα στο κουμπαρα και τα βαζουμε οσο το δυνατον πιο λιγα και απο την αλλη δεν δισταζουμε οταν υπαρχει μια ανάγκη που αναδύεται να ζητήσουμε από τον προπολογισμό της Ένωσης να ανοίξει ας πούμε και να καταβάλει ποσά. Ε, κατηγορούν το Κοινοβούλιο επίσης ότι είναι έτσι, σπάταλο, ενώ όχι, τα κράτη-μέλη. Το, συντομότερο, το συχνότερο είναι αυτό που συμβαίνει, να αποφασίζουν να, δαπαν, να δαπανίσουν και να βγάλουν λεφτά ας πούμε, από τον κουμπαρά για νέες δαπάνες. Δεν θα ξαναμιλήσω για το, το πώς επηρεάζουν οι κρίσεις στον προϋπολογισμό, παραδείγματος χάρη πολύ δηλαδή, για την ε, μετανάστευση, ας πούμε, και να χρηματοδοτήσουμε ε, την ε, μετεγκατάσταση αλλά και την εξωτερική διάσταση που ήταν πολύ υποτιμημένη στο ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Χρειάστηκε να, να εφεύρουμε νέους μηχανισμούς προϋπολογισμού. Ε, συνήθως η Κομισιόν έχει αυτό το καθήκον και για την κρίση των επενδύσεων όπως υπόθηκε έχουμε έλλειμμα 300 δις επενδύσεων α, κατέτος. Και το σχέδιο Juncker αναγκάστηκε να ψάξει να βρει στην έρευνα και στις υποδομές ε, των μεταφορών κάποια δισεκατομμύρια που δεν έβρισκε αλλού. Για την ανεργία των νέων είναι χειρότερα, γιατί η εγγύηση για την νεότητα που υπήρχε στο Πουδουπού 2014-2020 μέχρι το 2016 ας πούμε ήταν μόνο και μόνο λεφτά για μια πρώτη αξιολόγηση. Και το 2016 μετά εξαφανίστηκε τελώς. Και ο μηχανισμός που άρχισε να εμφανίζεται, να αναδύεται, ε, έχει υποστεί προσωρινή αναστολή. Σοβαρό. Τέλο πάνω. Πού βρισκόμαστε σήμερα και το λέω με μεγάλη σύνεση, γιατί προς το παρόν ε, τα συζητάει αυτά τα θέματα το Κοινοβούλιο. Σα δίνω διάφορα στοιχεία, έτσι, πάνω στα οποία δουλεύουμε κιόλας. Καταρχάς, η δομή του προπολογισμού, που είναι κάτι γνώμη μου ένα κεντρικό σημείο. Δηλαδή δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε ένα προπολογισμό που συντίθεται πάνω από το 80% του από τα τσεκ των κρατών μελών, γιατί αλλιώς ο μηχανισμός της ανταπόδοσης που θέλουν ορισμένα να εγγράψουν και στις συνθήκες θα πριτανεύσει αν παραμείνουμε σε αυτή την κατάσταση με τις επιταγές. Πρέπει να δουλέψουμε λοιπόν πάνω στην δομή του προπολογισμού της Ένωσης και όπως είπε και ο πρόεδρος αυτού, καλό είναι που πέφτει φέτος η έναρξη των εργασιών της Επιτροπής ε, Μόντι, της ομάδας υψηλού επίπεδου δηλαδή, που δουλεύει για το θέμα των ιδίων πόρων. Είναι μια ομάδα υψηλού επίπεδου που αποτελείται από ε, βουλευτές, από μέλη του Συμβουλίου και μέλη της Κομισιόν και προσπαθεί να βρει διέξοδο σε αυτό το αδιέξοδο που παραλύει την Ένωση. Αν όμως υπήρχε μία φορολογία με εισρωές προς τον ε, κοινοτικό προϋπολογισμό, η δουλειά των ε, Ευρωβουλευτών θα ήταν πάρα πολύ ζωτική σημασία. Γιατί η εισπραξη φόρων είναι η αρμοδιότητα των Εθνικών Κοινοβουλίων και επομένως ε, η συνεργασία με, τον Εθνικό Κοινοβουλ... με, τα... Εθνικά Κοινοβούλια θα ήταν εκ των Ουκάνευ. Και καλό θα ήταν να σκεφτούμε μαζί πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε αυτή τη δομή. Δεύτερον, να βελτιώσουμε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ένα από τα μείζωνα θέματα αυτό και που απορρέει από τις ίδιες ανάγκες και εδώ λοιπόν οι εθνικοί βουλευτές ε, θα έπρεπε να παίξουν κάποιο ρόλο γιατί το Συμβούλιο το οποίο παρεμβαίνει εδώ ο συνομοθέτης σύνομοθέτη αντί για τα εθνικά κοινοβούλια θα έλεγα για να το πω έτσι. Βλέπω ότι με κοιτάνε επίμονα. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Το θέμα της ενότητας του προπολογισμού. Με την κρίση των προσφύγων χρειάστηκε να εφεύρουμε ε, κάποιους ε, ε, δορυφορικούς προϋπολογισμούς, θα το πω έτσι, με πολλή φαντασία. Δημιουργεί πρόβλημα, γιατί, να και η δημοσιονομική ανηλικρίνεια, πού είναι ο δημοκρατικός έλεγχος, όλα αυτά τα, όλοι αυτοί οι δορυφορικοί ας θα πρέπει να επανεξεταστούν ε, καθώς θα γίνει αυτή η αναθεώρηση του πουδουπού. Και το θέμα τη διάρκεια βέβαια του πλαισίου. Γιατί. Ψηφίστηκε το 2013 το πλαίσιο, αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο και ξεκινάει το 2014. Ε, δημοκρατικός πώς είναι αμφισβητήσιμο. Και πάει μέχρι το 20. Δηλαδή, τη στιγμή που, ή μάλλον αυτοί που εξελέγησαν το 2014 ε, μπορεί να μην είναι ξανά το 2019. Δηλαδή, θα αποφασιστεί η δημοσιονομική κατάσταση, έχει αποφασιστεί πριν από αυτού, πριν από εμά που είμαστε τώρα εδώ, για μια ε, χρονική περίοδο που πάει που τους ξεπερνάει, λέει, θα, θα συνεχιστεί και μετά τη δική του θητεία. Υπάρχει ένα δημοκρατικό θέμα εδώ, ας πούμε, του προπολογισμού και της συναπόφαση από το εθνικό και τα, και το Ευρωπαϊ... εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν και κάποιες τεχνικές ε, ερωτήσεις, αλλά σημαντικέ θέμα τη ευελιξίας. Γιατί όπω υπόθηκε, η μερίδα του λέοντο του προπολογισμού της Ένωσης ε, ήδη είναι σαφές το που πηγαίνει. Ας πούμε τα, το Ταμείο Συνοχής. Δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε δηλαδή. Το θέμα είναι να δούμε τι ευελιξία μπορούμε να έχουμε λοιπόν από εκεί και πέρα. Και βέβαια το θέμα των οροφών, των των ορίων. Είμαστε σε θέση να αυξήσουμε τα, τις οροφές. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Σήμερα έχουμε κάποιες πολιτικές, παραδείγματος χάρη για τους πρόσφυγες, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για την ασφάλεια, για τα σύνορα. Γιατί αν το Σέγγεν διαλυθεί, ίσως γίνει αυτό γιατί τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχουν πραγματικά. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα θα πρέπει να τεθούν. Προφανώς δεν αφορούν μόνο τον προπολογισμό, αλλά πρέπει να τεθούν και να συζητηθούν. Εκεί φτάσαμε στις συζητήσει μας, αλλά για να ολοκληρώσω θέλω να σας πω και το εξή. Βασιζόμαστε στα Εθνικά Κοινοβούλια για να εργαστούμε Είμαστε και οι μεν και οι δε νόμιμοι φορείς για να εκπονήσουμε μια ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική και γι' αυτό μαζί θα πρέπει να γράψουμε αυτές τις σελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τώρα ανοίγουν μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος, για την παρουσίαση αυτή των ε, εργασιών της Επιτροπής Προϋπολογισμών σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Κόλμες, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Οικονομικών Θεμάτων της Βουλής Αντιπροσώπων στις κάτω χώρες. Και θέλω να πω στον κύριο Κούλμες ότι βασίζουμε πολλές ελπίδες στην Ολλανδική Προεδρία γιατί θα πρέπει να μας βοηθήσει να βρούμε την απαραίτητη ευκαμψία. Και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να λάβω εδώ το λόγο ενώπιόν σας. Θα ήθελα να παρουσιάσω την άποψη του Ολλανδικού Κοινοβουλίου για τα θέματα του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Το κόμμα μου, το D66 στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο, ίσως το πιο ευρωπαϊστικό κόμμα <clears throat> στο Κοινοβούλιο των κατοχωρών Αλλά ακόμα και εμείς και εγώ δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τον τωρινό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να γίνει μια συζήτηση των Εθνικών Κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το μέλλον των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών. Πριν από δύο εβδομάδε οργανώσαμε μια συνδιάσκεψη στο Άμστερνταμ για το μέλλον του προπολογισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ετήσι του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, γιατί είχαμε πολλέ επικρίσει τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τον προπολογισμό και τι διαδικασίε του. Ανησυχούμε για τι διαδικασίε που ακολουθούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε πεπισμένοι ότι είναι απαραίτητε οι μεταρρυθμίσει σε τρει τομεί. Πρώτον, <clears throat> είναι πολύπλοκο και απρόβλεπτο το σύστημα των εσόδων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, η λογοδοσία σε ό,τι αφορά τι δαπάνε. Και τρίτον, Χρειάζεται μεγαλύτερη ευκαμψία μέσα στις πολιετήσεις δημοσιονομικές προοπτικές και μεγαλύτερη εστίαση στην προθέμενη αξία των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα τρία θέματα λοιπόν θέλω να διαλάβω. Έσοδα. Από τότε που έγιναν οι διορθώσεις στον προπολογισμό του 2014, εμείς ακόμα προσπαθούμε να βρούμε άκρη με τον κύριο Ντάσελμπλουμ, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών γιατί το σύστημα αυτό είναι απρόβλεπτο, χρειάζονται επαναυπολογισμοί επί τη βάση του ΑΕΧ και χρειάζονται συνεχείς διορθώσεις. Θα ήταν πολύ καλό να μπορέσουν να γίνουν με σταθερές, σε σταθερές χρονικές στιγμές οι διορθώσεις και οι υπολογισμοί. Αυτό θα κάνει πιο εύκολο το εθνικό έργο. Κοιτάμε επίσης τι γίνεται με την ομάδα υψηλού επίπεδου του κυρίου Μόντι για του ίδιου πόρου, αλλά θέλουμε να θαρρύνουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλία και τα Εθνικά Κοινοβούλια να εξετάσουν τι ενδεχόμενε μεταρρυθμίσει για τα έσοδα, ώστε να υπάρχει ένα σαφέ και αποτελεσματικό σύστημα σύλλογη εσόδων για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Δεύτερο θέμα, το θέμα των δαπανών μα. Λέει το ελεκτικό συνέδριο εδώ και 20 χρόνια, κάθε χρόνο, ότι δεν δαπανώνται σωστά τα λεφτά των φορολογουμένων. Και αυτό σημαίνει ότι σκάβει τον ίδιο τον τάφο της η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί οδηγεί σε όλο και πιο μεγάλη δυσφορία που είναι όλο και πιο έντονη από τους πολίτες. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δέκα χρόνια, οι κάτω χώρες έχουν κάνει μια εθνική δήλωση αξιοπιστίας σε ό,τι αφορά τα ποσά που δαπανάει η Ολλανδική κυβέρνηση, τα ευρωπαϊκά κονδύλια που δαπανά στις κάτω χώρες. Πιστεύουμε ότι για να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία θα πρέπει τα κράτη-μέρη τουλάχιστον να δημοσιεύουν μια εθνική δήλωση κάθε χρόνο. Το τρίτο θέμα μου είναι περισσότερη ευκαμψία και προσθέμενη αξία. Έχει ενώπιον τη τεράστιε προκλήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οικονομική κρίση και την κρίση των προσφύγων, αλλά το μισό προπολογισμό τη η Ευρωπαϊκή Ένωση τον δαπανά στις, στις προτεραιότητες του χθες και όχι σε αυτές του σήμερα και όχι του αύριο. Ο προπολογισμό λοιπόν δεν πρέπει να παραμένει άκαμπτος για κάθε 7 ετία, αλλά θα πρέπει να προσαρμόζεται στι ανάγκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, οι δημοσιονομικέ προοπτικέ τη πολιετή θα πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται με μεγαλύτερη ευελιξία, να υπάρχουν μεταφορέ μεταξύ κεφαλαίων για να μπορεί να είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε σε νέε πολιτικέ και οικονομικέ προκλήσει. Πέραν τη ευκαμψία και ευελιξία, μια πλειοψηφία των βουλευτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Ολλανδία θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή για την διατύπωση συγκεκριμένων στόχων για τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ο ιδανικό προπολογισμό θα πρέπει να εξυπηρετεί στόχου οι οποίοι πραγματικά προσφέρουν προσθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προστασία των εξωτερικών ε, συνόρων, ασφάλεια, βιώσιμη ενέργεια, και καινοτομία. Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά από μεμονωμένα κράτη-μέλη. Η επιλογή των ε, σχεδίων θα πρέπει να γίνεται επί τη βάση προσθέμενης αξίας και όχι επί τη βάση εθνικών προτεραιοτήτων. Εν κατακλείδου. Είμαστε ιδιαίτερα αδίμονες να ακούσουμε από τα άλλα κρατημέλη και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ποιε είναι οι ενέργειες που έχουν γίνει για να γίνει πιο ευέλικτος ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και πιο αποτελεσματικός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κόλμες. Καλώς. Έχοντας ακούσει τους δύο εισηγητές μας, νομίζω τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Πρώτος ο μιλητής είναι ο Φρανσούα Μάρκ, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της Γαλλικής Γερουσίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έχουν λάβει το λόγο προηγουμένως και για τις ε, λεπτομέρειες που μας έχουν δώσει, για το ανοιχτό πνεύμα που έχουν παρουσιάσει, την κυρία Τόμα και τον κύριο Κόλ μες σε σχέση με την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα του προϋπολογισμού. Και εγώ από τη δική μου πλευρά <clears throat> πιστεύω ότι η ευελιξία στη χρήση των κονδυλίων του προϋπολογισμού χρειάζεται βελτίωση. Είναι και μία από τις κατευθύνσεις που έχει αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την πρόταση που θα διατυπώσει στα μέσα του 2017 και ελπίζω ότι θα μπορέσει να υλοποιηθεί για μια καλύτερη στόχευση των κονδυλίων και την διευκόλυνση για τη χρήση καινοτόμων χρηματοοικονομικών εργαλείων. Όλα αυτά λοιπόν είναι <clears throat> θετικά και επιθυμητά και πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή το ταχύτερο δυνατόν. Θα ήθελα τώρα να διευκρινίσω ότι σήμερα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 74% των δαπανών πηγαίνουν στην γεωργία και στο περιβάλλον 40% και στην πολιτική συνοχής κατά 33%. Επομένως τα δύο αυτά μεγάλα κεφάλαια θα πρέπει να εφαρμόσουν ήδη την ευκαμψία και την ευελιξία. Αλλά αυτό δεν φαίνεται να γίνεται. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει το ερώτημα αν μπορούμε να έχουμε μια αποτελεσματική αλληλεγγύη με τους ε, πρόσφυγες και αυτό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στην πολιτική συνοχή. Μας είπε σήμερα το πρωί ένα Έλληνα βουλευτή ότι η χώρα του χρειάζεται να πληρώσει την ύφη σε ύψο ενό δισεκατομμυρίου και ζήτησε τη βοήθεια τη Ευρώπη για να καλύψει τι δαπάνε για του πρόσφυγε. Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι προπολογισμοί μα μπορούν να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα. Δεν μιλάμε τώρα να δημιουργήσουμε νέα φορολογικά μέσα, νέου φόρου και ούτε και οι πολίτε μα το θέλουν. Κανεί δεν θέλει να έχει νέου φόρου. Αλλά μήπω μπορούμε να κατευθύνουμε ορισμένε δαπάνε του προπολογισμού μα προ τι ε, επιτακτικέ ανάγκε που ε, αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και όχι στη Γεωργία. βλέπουμε σήμερα στην ε, Ευρώπη, έτσι όπως είναι οργανωμένη η χρηματοδότηση της γεωργίας, να μην μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά θα πρέπει να το θέσουμε το θέμα αυτό σε επίπεδο προϋπολογισμών. Γιατί η φιλελεύθερη, φιλελεύθερη πολιτική η οποία έχει ακολουθήσει θεωρεί ότι η αγορά θα τα λύσει όλα και έχει περιστύλει τους πόρους που είναι διαθέσιμοι από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η πολιτική αυτή στη Γεωργία απέτυχε η πολιτική για την κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων απέτυχε. Και εκεί η Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να διορθώσει την πορεία της και το ερώτημα είναι αν μπορούμε λοιπόν <clears throat> στον τομέα της συνοχής και στον τομέα της γεωργίας να έχουμε μια πραγματική ευελιξία. Χωρίς μικρόφωνο ο Ευχαριστώ. Είναι καλό που έχουμε ανθρώπους εκλεγμένους, αιρετούς εκπροσώπους από διάφορες χώρες της ε, Βρυξέλλες. Οι τρέχουσες δημοσιονομικές ε, πολιτικές ε, γεννήθηκαν ε, όχι σε μια εποχή κρίσης και δημοσιονομικής εξυγίανσης. Έχουμε τώρα την επιπλέον πίεση του κυρίου Κάμερον που ασχολείται και με άλλα θέματα αλλά και ε, για το θέμα του προϋπολογισμού. Και τώρα πρέπει για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε μειωμένο προϋπολογισμό με μεγαλύτερη ευελιξία. Ταυτόχρονα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον είναι μονόδρομος ε, το σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει. Σύμφωνα με την συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε νέες ε, πολιτικές που πρέπει να χρηματοδοτούνται, το διάστημα, την κλιματολογική αλλαγή. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα χρήματα. Αυτά ε, και οι προκλήσεις της μετανάστευσης είναι η νέα μας πραγματικότητα. Είμαστε στην αρχή του 2016. Η κατάσταση τώρα είναι λίγο παραπλανητική γιατί έχουμε αυτό το, αυτή τη μεγάλη στέρηση στις πληρωμές που έχουν συσσωρευτεί και αυτό έρχεται να, να συνδυαστεί με νέα προβλήματα. Πρέπει λοιπόν αυτό το βουνό των ε, μη πραγματοποιηθήσεων πληρωμών να αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα με τις νέες ε, δυσκολίες που έχουμε τώρα και αυτές που θα έρθουν τα επόμενα χρόνια. Έχουμε ήδη εξ το 2016, έχει κινητοποιηθεί το εργαλείο ευελιξίας, έχει γίνει μεγάλη ε, χρήση της εμπροστοβαρούς φύσης του προϋπολογισμού. Χρησιμοποιηθήκαν χρήματα ήδη που πρέπει να πληρωθούν το 18, 19 και 20. Είναι αυτό το περιθώριο για τις έκτακτες ανάγκες που έχουμε, με άλλα λόγια. Άρα ε, τώρα δεν είμαστε απλώς σε μια φάση αναθεώρησης και επανεξέτασης, αλλά σε μια φάση σοβαρής επανεξέτασης για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις ε, καθώς έχουμε μείνει με τόσους απλήρωτους λογαριασμούς βάση του πλαισίου του 14. Ε, επίσης υπάρχει το θέμα των οραφών. Υπάρχει το θέμα της μετανάστευσης, η διεθνής ευθύνες, το νέο μάντρα της προστιθέμενης αξίας δεν θα μας βοηθήσει και πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν διάφοροι ορισμοί της προστιθέμενης αξίας. Μπορεί να είναι και οι τοπικές επενδύσεις και η καινοτομία για την ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά, ε, ίσως ε, και το θέμα των ΣΔΙΤ να μας απασχολήσει, που είναι λίγο πιο πολύ ε, μια νοοτροπία των βόρειων χωρών, δεν είναι ένα θαυματουργό όπλο, ε, οπότε σίγουρα χρειαζόμαστε μια μεγάλη αναθεώρηση. Ευχαριστούμε τον κύριο Λεβαντόφσκι. Γιάννη Μυριάντα έχει το λόγο. Χαιρετίζουμε αυτή τη διαδικασία αναθεώρησης του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ, αλλά πρέπει να είμαστε στρατηγικοί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και σε επίπεδο Εθνικών Κοινοβουλίων. Γιατί πολλά διακυβεύονται και αν όντω ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συμπληρώσει τι προσπάθειε που κάνουν τα κράτη σε εθνικό επίπεδο, δεν πρέπει να αντιδρούμε απλώ σε αυτά που συμβαίνουν. Πρέπει να είμαστε πιο προμηθείς. Ε, τώρα, με μία μείωση 85 δι. σε σχέση με το προηγούμενο πι, το νέο πι πρέπει να χρησιμοποιήσει νέα εργαλεία και νέες ε, δομές. Έχουμε συστηματικά καθυστερημένες πληρωμές για τα προγράμματα 2014-2020, ειδικά αυτά που προωθούν την ανάπτυξη, την κοινωνική και ε, δημόσια επένδυση ειδικά για την νεολαία. Το ίδιο ισχύει και για τις ανάγκες των προσφύγων. Έτσι λοιπόν τώρα έχουμε την ευκαιρία αυτής της αναθεώρησης ε, να είμαστε γενναίοι και υπεύθυνοι και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις έκτακτες ανάγκες και τις προκλήσεις. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα των εσόδων. Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι η Κομισιόν έχει τον κατάλληλο χρόνο και τους δέοντες πόρους για να καταβάλει τις πληρωμές στα κράτη-μέλη. Ε, Ποιε είναι οι προτάσεις που κατατίθενται για να αντιμετωπίσουμε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε, για τους ε, ωφελούμενους του Λίντερ στην Ιρλανδία. Ξέρω ότι ακόμα περιμένουν τις πληρωμές τους και το ίδιο ισχύει και σε άλλες χώρες. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε το θέμα των δαπανών. Θα ήταν καλύτερα λοιπόν να, μιλω, να μιλήσουμε περισσότερο για την ενότητα του προϋπολογισμού, να μην έχουμε ad hoc δομές, να βελτιώσουμε επίσης τη λογοδοσία σε επίπεδο προϋπολογισμού, ενώ ενισχύουμε τον δημοκρατικό έλεγχο για να διασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτούνται μέσω και από τον προϋπολογισμό. Τι έχετε να πείτε σε σχέση με αυτό. Ευχαριστώ ο Βλαδιμίρ Μάγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι ακούμε μέχρι τώρα, η πλειοψηφία από εμά θα μπορούσε να συμφωνήσουν ότι χρειάζονται κάτι, καλύτεροι κανόνες για τις πληρωμές από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνούμε όλοι ότι οι πληρωμές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για σχέδια τα οποία προσθέτουν σε προσθεμένη αξία για το ευρωπαϊκό επίπεδο και βοηθούν και την απασχόληση. Ξέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού ξαναγυρίζει στα κράτη-μέλη. Το πρόβλημα για μένα βρίσκεται στους ίδιους πόρους. Στην τελευταία διακοινοβουλευτική συνάντησή μας υπήρξαν μέλη από τα Εθνικά Κοινοβούλια της Γαλλίας και της Ισπανίας που μας λέγανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αθυστερούμενα για πάρα πολλά χρόνια και τα κράτη δεν δίνουν λεφτά για να καλύψουν αυτά τα χρωστούμενα και σε τοπικό επίπεδο οι δήμαρχοι διαμαρτύρονται ότι δεν πληρώνονται τα λεφτά που έχουν καταβάλει στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε συμμάχους για να υπάρξει πίεση για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Είναι δύσκολο να έχουμε συμφωνία με το Συμβουλή. Γι' αυτό χρειαζόμαστε εσά, τα Εθνικά Κοινοβούλια, ω σύμμαχου για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Ξέρουμε ότι τρίτε χώρε όπω η Κίνα και άλλε χώρε εξάγουν αγαθά προ εμά, τα οποία παραγόνται με τρόπου οι οποίοι είναι εχθρικοί για το περιβάλλον. Γιατί να μην φορολογούνται όμω αυτά τα αγαθά στα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το ίχνος διοξιδίου του Άνθρακο που έχει να κάνει με την Παρασκευή τους. Επομένως αγαπητοί φίλοι, αν έπρεπε να συνοψίσω, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει εμεί να διατυπώσουμε ιδέες και μετά η ομάδα του κυρίου Μόντι να πιέσει τα κρατη να καταλήξουμε σε μια λύση γιατί το Σαντουσκό δεν είναι πια αποδεκτό. Ευχαριστώ λέω ο Ο κύριος Μάκα είναι από την Σοσιαλιστική Ομάδα και τη Σλοβακία. Η Άιντερ Κουάρδια Σαβάλ η οποία είναι Γενική Εισηγήτρια του Προεπορισμού για το 2016, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η οποία είναι εκλεγμένη φυσικά στην Ισπανία. Και εκπροσωπεί όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ζήτησα το λόγο όταν ε, μίλησε ο κύριος Κόλμες αναφέρθηκε σε τρία κομβικά θέματα για το δημοσιομικό πλαίσιο και μου έκανε μεγάλη εντύπωση το τρίτο σημείο που ανέφερε που είχε να κάνει με την, με ακούτε, με την ευελιξία. Προστέμενη αξία ευρωπαϊκή και ευελιξία. Και για το θέμα της ευρωπαϊκής προστέμενης αξίας, ήδη αυτό είναι ένα επίμαχο θέμα γιατί ο καθένας έχει μια διαφορετική εκτίμηση για το τι σημαίνει αυτό, αλλά για την ευελιξία. Στην συνδιάσκεψη που οργανώσατε η Ολλανδική Προεδρία και εγώ ήμουν σε αυτή την ομάδα εργασία που μιλήσαμε για την ευελιξία. Και δεν καταφέραμε ούτε εκεί να καθορίσουμε τι είναι η ευελιξία και πέραν του τι είναι, πώς θα την εφαρμόσουμε. Α είμαστε ειλικρινέ, Με ένα προπολογισμό του 1% του ΑΕΠ τη Ευρωπαϊκής ένωση όπου κάθε φορά που υπάρχει μια κρίση βλέπουμε τον προπολογισμό σαν να είναι αγελά για άρμεγμα και αν είναι η λύση για να ε, καλύψουμε τα προβλήματα, προφανώς δεν υπάρχει χρήμα για τίποτα άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν. Μπορεί κανείς να μιλήσει για τις παλιές προτεραιότητες και τις νέες προτεραιότητες. Κανείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε και στα Εθνικά Κοινοβούλια αρνείται το γεγονός ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί ο Ευρωπαϊκός προπολογισμό, να γίνει μελλοντόστροφος, να μπει σε πολιτικές όπως είναι η τεχνολογία, η καινοτομία, ο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Νομίζω ότι εκεί συμφωνούμε και Εθνική και ε, Ευρωπαίοι βουλευτέ. Το θέμα είναι πώς θα, πού θα βρούμε τα χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε αυτέ τι νέε πολιτικέ. <clears throat> θα οδηγήσουμε σε παράθεση των παλαιών προτεραιοτήτων με τι νέε προτεραιότητε. Είναι αλήθεια ότι η γεωργία και η συνοχή καλύπτουν το 74% του προπολογισμού. Αλλά σίγουρα αν μπορούμε να, να βελτιώσουμε τα προγράμματα τη συνοχή και τη γεωργία είναι απαραίτητο να διατηρηθούν αυτά. Είναι απαραίτητο να έχουμε διαφορετικά ταμεία και ταμεία συνοχή για να βοηθήσουμε τι πιο φτωχέ χώρε. Είναι απαραίτητο να έχουμε στήριξη για του γεωργού. Πώ λοιπόν θα χρηματοδοτήσουμε τι νέε πολιτικέ, ή θα βρούμε περισσότερα χρήματα, ή αλλιώ θα στρέψουμε μερικέ προτεραιότητε έναντι των άλλων. <clears throat> Αυτό λοιπόν είναι μια γενικότερη συζήτηση που δεν αφορά μονάχα την ενδιάμεση αναθεώρηση, αφορά και τις επόμενες, το επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψη τη Ολλανδική Προεδρίας σχετικά με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντόγκε, που είναι Γερμανός ε, βουλευτής, μέλος της ομάδας του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα την παρουσίαση του κυρίου Κρόμες και επιτρέψτε μου κάποιες, ε, κάποια κριτική. Ε, αναφερ, αναφερθήκατε στη δήλωση αξιοπιστίας που χρησιμοποιείται από το ελεγκτικό συνέδριο. Έχουμε το 80% λοιπόν του προϋπολογισμού που πρέπει να διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Είναι τα διαρθρωτικά ταμεία και η γεωργική πολιτική. Ε, και το ελεγκτικό συνεδρίο πάντοτε επικρίνει τον τρόπο εφαρμογής του προϋπολογισμού. Το 2013 όταν ε, με τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο ε, Λεβαντόφσκι και τον κύριο Γιάν Μόλτερ από την Ολλανδία έκανα μία έκθεση για το θέμα. Είδα ότι τα κράτη-μέλη αρνούνταν να υπογράψουν δήλωση αξιοπιστίας για τα κονδύλια που χρησιμοποιούν οι χώρες τους από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι θεωρώ πως είναι καλό το γεγονός ότι, ότι συζητούμε αυτά τα θέματα εδώ και όπως ε, το Νοέμβρη συζητήσαμε με την Επίτροπο Γεωργίευα στην Επιτροπή φυσικά πρέπει να γίνει η συζήτηση για την προστιθέμενη αξία. Ποιε είναι οι δαπάνες που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ποια είναι η προστιθέμενη αξία που έχουν αυτές. Αυτό είναι μία από τις τρέχουσες προκλήσεις ε, ε, λόγω των εξελίξεων ε, που γίνονται όλο και πιο επίγουσες. Μιλάμε για περισσότερη ευελιξία επίσης. Το μήνυμα είναι σωστό, αλλά ε, μου λείπει η πίστη. Ποιος ε, όποιος προσπαθήσει να φέρει περισσότερη ευελιξία ε, στις προσπάθειές μας, όπως έγινε και στο προηγούμενο πι όπως γίνεται ε, και όπως έγινε την τελευταία στιγμή το, στο πι 2014-2020 που, που έγιναν προσπάθειες πλοκαρίσματος, ε, αυτά προέρχονται όλα από τα κράτη-μέλη. Αν το Κοινοβούλιο τελικά ε, δεν είχε ε, ε, συμβουλέψει κάποια πράγματα για το τρέχον πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, τώρα θα είχαν τελειώσει τα οικονομικά, γιατί η δική μας ευελιξία αυτή που εμείς διαπραγματευτήκαμε χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του νέου πακέτου των Δύση για τους πρόσφυγες, το οποίο μπορέσαμε να θεσπίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ήταν 9,2 έτσι λοιπόν, στην τελευταία ανάγνωση, το καλοκαίρι στην Κορεπέρ, έγινε ακόμη μια προσπάθεια να ε, σταματήσει πλήρως η τρέχουσα αυτή η προσπάθεια και εξέλιξη. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το επίπεδο και τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά και η πολιτική των κρατών μελών, εξ αρχής να αναλάβουν την ευθύνη τους ε, για τις διαπραγματεύσεις και τα αποτελέσματα, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα που από κοινού τώρα ξεκάθαρα υποστηρίζουμε και ούτε θα είχαμε κάνει αυτές τις προόδους που ε, κάναμε και ήταν απαραίτητες. Και τώρα αυτό που βιώνουμε είναι να έχουμε τη δημιουργία νέων ε, χρηματοοικονομικών μέσων, νέων ε, projects, νέα προγράμματα, τα οποία όμως είναι εις των μεταφορών και της έρευνας. Βέβαια, ε, σε αυτή την πρώτη φάση ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν κινηθεί, αλλά πρέπει να γίνει και η τελευταία αξιολόγηση. Τώρα για την ευελιξία, λόγω της απλούστευσης ή λόγω του ότι αποφεύγεται η αναθεώρηση ε, στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, φαίνεται ότι κόβονται τα προγράμματα γειτονίας ή αλλάζουν η μορφή τους, όπως ας πούμε αυτά για την Αφρική και περιμένουμε τα κράτη-μέλη να, κάνουν, ε, να δώσουν τη συμβολή τους ε, αντίστοιχα. Είναι αυτό μια δοκιμή για να δούμε αν αυτά τα μέσα θα λειτουργήσουν ή αν θα πρέπει να τα ε, σταματήσουμε. Και μια τελευταία παρατήρηση, η οποία έχει να κάνει και με την επόμενη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε. Αυτό που κάναμε ε, στις αρχές Οκτωβρίου μαζί, ε, από κοινού δηλαδή και με θάρρος, ε, έκανε ξεκάθαρο δύο κατηγορίες συγκεκριμένα να μην μπορούν πλέον σε επίπεδο προϋπολογισμού να αντιμετωπίσουν τα πράγματα που έχουν στη μερίσια διάταξή τους. Η προστασία των συνόρων, το θέμα της Frontex το θέμα του αν θέλουμε ουσιαστικά να έχουμε ε, νέα βήματα στα προγράμματα γειτονίες και να συμβάλλουμε ώστε το περιβάλλον γύρω μας ε, να είναι σταθερό ή στην ουσία ε, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα απαντήσουμε κατά την αναθεώρηση σε αυτές τις νέες ερωτήσεις δεν έχουμε απαντήσεις και ε, μιλάμε για τα διαρθρωτικά ταμεία και την κοινή γεωργική πολιτική και όποτε φύγουμε αυτό το θέμα φύγονται κάποια κράτη-μέλη. Όποτε και να γίνει αυτό, ε, στην ουσία καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να βρούμε κάποια κονδύλια τα οποία μπορούν να αλλάξουν προορισμό και να αντιμετωπίσουμε τις ε, έκτακτες ανάγκες. Ευχαριστούμε πολύ ακόμα και για την αναφορά σας στην επόμενη συζήτηση, λέει ο Πρόεδρος. Δεν πρέπει να έχουμε πολλές ε, ε, προσδοκίες για το πώς θα προχωρήσουν τα θέματα του προϋπολογισμού. Τώρα, ε, ως εκπρόσωπος, μάλλον ως εκλεγμένο μέλος από την Εσθονία και μέλος της Επιτροπής του Προϋπολογισμού και των Πρασίνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριο Στάραντ. Με ενδιέφερε η, παρουσία, παρουσίαση του Ολλανδού εκπροσώπου που μίλησε για τρία δημοσιονομικά προβλήματα. Μεγαλύτερη ευελιξία, το άλλο είναι το να τη ζητάμε και άλλο να τη δίνουμε. Προς το παρόν, η καλύτερη λύση βρίσκεται στα χέρια των εθνικών βουλευτών. Γιατί μόνο εκείνοι μπορούν να εξαναγκάσουν τις κυβερνήσεις τους να συμφωνήσουν ότι μια ενδελεχής αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Αλλιώς τα προβλήματα ακαμψίας θα συνεχίσουν να μας ταλανίζουν. Μόνο τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να αναγκάσουν τις κυβερνήσεις τους να το κάνουν αυτό. Εμείς από εδώ δεν μπορούμε. Και αν το Συμβούλιο δεν κουνηθεί, αν δεν χαλαρώσει την τον ασφικτικό εναγκαλισμό που ασκεί στην Κομισιόν δεν μπορούμε να μιλάμε για αναθεώρηση. Και με βάση τη συνθήκη ε, εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να τους εξαναγκάσουμε με την ψήφο μας να κάνουν κάτι που δεν θέλουν και θέλουμε εμείς. Επομένω τίποτα θα γίνει. Όταν όμως τα μέλη του Συμβουλίου αισθανθούν αυτή την κάψα της κολάσεως στο σβέρκο τους, το, την ανάσα αυτή θα την στέλνουν οι εθνικοί βουλευτές, τότε μπορεί η κατάσταση να αλλάξει και να έχουμε μια ουσιαστική αναθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού πλασίου. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ. Ο κ. Καριέλο Φραντσέσκο από την Ιταλία, μέλος του, της Ιταλικής Βουλής στη Ρώμη. Ευχαριστώ, ο κ. Καριέλο. Θέλω να αξιολογήσουμε σε ποιο βαθμό η δουλειά της διαθεσμικής ομάδας που είχε σαν στόχο να αξιολογήσει τους δείκτες επίδοσης για τη χρήση των διαφόρων κοινοτικών ταμείων γίνεται σωστά. Για να δείξει στους Ευρωπαίους πολίτες τι χρήση γίνεται των κοινοτικών ταμείων ε, και των κονδυλίων που παίρνουν τα διάφορα κράτη-μέλη και κατά πόσον ε, επενδύουν πραγματικά στην κοινότητα αντί να ξοδεύουν τα λεφτά αυτά για πάρτι τους, για να το πούμε έτσι. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η ομάδα εργασίας να δείξει στους Ευρωπαίους πολίτες για να τους αποδείξει ότι αξίζει τον κόπο να επενδύουμε και να δίνουμε λεφτά στα ευρωπαϊκά ταμεία και από εκεί να τα χρησιμοποιούμε. Αν έχουμε αντικειμενικά κριτήρια για κάθε επένδυση κοινοτική και αν ε, η συγκεκριμένη επένδυση δεν ε, βοηθάει στην ε, αναθεώρηση, δεν, βοηθάει στην ανάπτυξη ολόκληρης κοινότητας, θα πρέπει να αναθεωρηθεί στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και να πάψει να υπάρχει συγκεκριμένη ας επένδυση. Διερωτώ με, έχει γίνει πραγματικά αυτή η δουλειά από την ομάδα μέχρι στιγμής. Αν έχει, έχει δώσει αποτελέσματα. Και αν ναι, θα πρέπει να δοθούν αυτά τα αποτελέσματα και στην Κομισιόν. Ευχαριστώ. Εδώ τα εθνικά κοινοβούλια θα μπορούσαν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Δηλαδή να αξιολογήσουν την, τη θετική επίπτωση των ευρωπαϊκών πιστώσεων. Και αν είμαστε σίγουροι ότι συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και στην ε, απασχόληση που είναι οι απόλυτες προτεραιότητες. Ή, επειδή υπάρχουν ευρωπαϊκές επενδύσεις και κονδύλια, κάνουμε επενδύσεις που δεν ε, ανταποκρίνονται στις προτεραιότητές μας. Δηλαδή, δεν έχουν να χρηματοδοτήσουν τις πραγματικές προτεραιότητές μας. Θα μπορούσε θα μπορούσε να ασκηθεί αυτό ο έλεγχο για τη χρήση που κάνουμε των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Τα, κοινοβούλια θα μπορούσαν να κάνουν αυτό το, αυτόν τον έλεγχο. Ε, Επίση, τονίζεται τη σημασία τη ευελιξία για τα απλήρωτα. Μέχρι στιγμή πάνε κάπω καλύτερα τα πράγματα. Γιατί τα προγράμματα του που, του 14-20 έχουν αναβληθεί λόγω τη περιπλοκότητά του για να διευκολύνουμε τι πληρωμέ. Έχουν ανασταλεί, α πούμε. Γι' αυτό έχουμε μια για, έχουμε μια προσωρινή ανακούφιση. Αλλά για το 17, 18, 19, 20 προβλέπουμε κόλαση. Γιατί έχουμε 24, είχαμε 24 δισεκατομμύρια απλήρωτων λογαριασμού στο τέλος του 2014. Παρακαλώ. Θα ήθελα... Κοιτάξτε, καταρχάς η Ολλανδία έκανε μια πρωτοβουλία οργανώντας μια διάσκεψη για το θέμα αυτό. Είδατε ότι τα νέα εργαλεία, η έννοια της προστιθέμενης αξίας ε, γύρει διάφορα ερωτηματικά. Το είδατε αυτό στην ε, σύνοδο αυτή. Αλλά αυτά τα ερωτηματικά θα πρέπει να τα απαντήσουμε. Ο κύριος Κούλβες έχει το λόγο για να απαντήσει τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Ως μέλος ενός Εθνικού Κοινοβουλίου πρώτα απ' όλα. <clears throat> Πάντα γνωρίζω ότι υπάρχει έλλειψη χρημάτων τα τελευταία 5,5 χρόνια στις κάτω χώρες εμείς μειώσαμε τις δαπάνες μας κατά 50 δισεκατομμύρια, 8% του ΑΕΠ και στην χώρα μας. Έχουμε πάντα συζητήσεις για την έλλειψη χρημάτων και τις καλές προθέσεις οι οποίες δεν αντανακλώνται σε επαρκή κονδύλια. Πάντα θα υπάρχει λοιπόν αυτή η συζήτηση για τα απαραίτητα κονδύλια. Και μετά υπάρχει αυτή η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί έχετε αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο το επτάετες, το οποίο είναι ουσιαστικά παγιωμένο και μετά τίθεται η συζήτηση για την ευελιξία. Γι' αυτό το Ολλανδικό Κοινοβούλιο έχει αυτή την ιδέα, προτού γίνει η διάμεση αναθεώρηση, να διοργανώσει ως Προεδρία του Συμβουλίου αυτό το συνέδριο στο Άμστερνταμ. Ξέρω και καταλαβαίνω ότι η προσθέμενη αξία είναι ένα δύσκολο θέμα γιατί διαφέρει από χώρα σε χώρα η αντίληψή ένα παράδειγμα, όταν εμείς στις κατοχώρες χρηματοδοτούμε ποδηλατόδρομους με ευρωπαϊκά χρήματα, νομίζω ότι είναι καλή λύση. Είναι χρήσιμη. Νομίζω είπε το αντίθετο. <laughs> και υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα. Μίλησατε επίση και για μια εθνική δήλωση αξιοπιστία. Από ό,τι ξέρω, μόναχα τρει χώρε τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουν <clears throat> διατυπώσει μια εθνική δήλωση αξιοπιστία και τα άλλα κράτη ποτέ. Και πράγματι έχετε δίκιο, 80% των χρημάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του προπολογισμού δαπανούνται από τι εθνικέ κυβερνήσεις οι οποίε πρέπει να απομιστούν την ευθύνη και να λογοδοτήσουν για αυτέ τι δαπάνε. Στον Ολλανδικό τύπο κάθε φορά που έρχεται η ετήσια έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου λένε οι Εφημερίδε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει λεφτά που πανεστράφει. Επομένω, είναι και ευθύνη των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει αυτή η εθνική δηλώση αξιοπιστία. Είναι θέματα που μπορούμε να συζητάμε βέβαια για ώρε. Ευχαριστώ. Λέω πρόεδρο, <clears throat> μα μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δαπανά τα λεφτά όπω να είναι. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά, αυτά τα οποία κάνουν ό,τι θέλουν με τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να καταδείξουμε είναι ότι έχουμε χρήματα που πηγαίνουν από τα κράτη-μέλη, πηγαίνουν στις Βρυξέλλες και ξαναγυρίζουν στα κράτη-μέλη, έχει νόημα αυτή η διαδικασία, έχει προσθέμενη αξία. Εάν λοιπόν αυτά τα χρήματα από την Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό δεν προκαλούν δημόσιες δαπάνες και γενικά παραγωγικό έργο, υπάρχουν και κράτη-μέλη τα οποία ουσιαστικά για να χρησιμοποιήσουν αυτά τα, αυτά τα κονδύλια αναγκάζονται να συνάπτουν χρέος. Λοιπόν, Πρόεδρε, ο κύριο Κόλμες προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Θα αντιδράσω κι εγώ. Πρώτον, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και το λέω σε όλους τους εθνικούς βουλευτές. Η συζήτηση να μην είναι μόνο το μελλοντικό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά και η αναθεώρηση του τρέχοντος. Ε, μου, με εντυπωσίασε πηγαίνοντα στο Άμστερνταμ και νομίζω ότι και όλοι οι Ευρω, ευρωβουλευτέ εντυπωσιάστηκαν πηγαίνοντα στο Άμστερνταμ ότι συζητούσαμε μόνο ε, για την επόμενη περίοδο, 2020 και μετά. Αλλά δεν μιλούσαμε για την αναθεώρηση του τρέχοντο. Έπειτα, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κόλμε στο επόμενο. Για το θέμα των, α, ε, της αδιαφάνειας των εσόδων. Ε, έχουμε και τους ε, ευρωπαϊκούς ε, βουλευτές και τους ε, εθνικούς βουλευτές οι οποίοι ας πούμε μερικές φορές δεν βλέπουν τις μυστικές συμφωνίες. συμφωνώ ότι υπάρχει αδιαφάνεια. Ε, επίσης, χρειάζεται ευελιξία, όπως είπε και η Ισπανίδα βουλευτής, το θέλει το Κοινοβούλιο, αλλά δεν θα λύσει το πρόβλημα του μικρού προϋπολογισμού. Όσο... Τι να σας κάνει τώρα η ευελιξία όταν ο προϋπολογισμός είναι τόσο στενός, ας πούμε. Βγάζετε από τη μια τσέπη για να βάλετε στην άλλη, ας πούμε. Εντάξει, όλα αυτά ναι, ευελιξία ναι, αλλά να είναι επαρκής ο προϋπολογισμός. Αυτό έγινε με το Ταμείο των Επενδύσεων και με την έρευνα και τις υποδομές. Για το θέμα της ε, προσθέμενης αξίας το ίδιο πράγμα είναι. Ίσως συμφωνούμε όλοι μας ότι θα πρέπει να δούμε α, αν υπάρχει προστιθέμενη αξία και να υπάρχει προστιθέμενη αξία. Αλλά αν είναι προτεραιότητα της Ένωσης ότι πρέπει ας πούμε να εγκαταλείψουμε ας πούμε το αυτοκίνητο, να, να τα σταματήσουμε να το χρησιμοποιούμε τόσο πολύ λόγω του ότι παράγει διοξείδιο του άνθρακα και θα πρέπει να έχουμε μια ήπια ανάπτυξη. Επομένως, το θέμα δεν είναι ο ποδηλατόδρομος στο χωριό μου ας πούμε, αλλά το θέμα είναι να έχουμε ήπια μέσα μεταφοράς παντού που από κοινού θα βελτιώσουν το περιβάλλον, την υγεία των Ευρωπαίων. Έτσι. Να η προστιθέμενη αξία εδώ. Εντάξει, επειδή μιλήσατε για ποδηλατόδρομους μιλάω κι εγώ γι' αυτό, έτσι. Ε, συγγνώμη τώρα, έτσι. Παρακαλώ, παρακαλώ να παρέμβετε. Ε, κοιτάξτε, η παρατήρησή μου δεν αφορούσε τη σημασία των ποδηλατόδρομων, αλλά τη χρηματοδότηση των ποδηλατόδρομων μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Είναι εθνική ευθύνη, ειδικά στην Ολλανδία. Δηλαδή η Ευρώπη καθορίζει μια προτεραιότητα. Υπέρ, τον ποδηλατόδρομο, χωρίς όμως οι ποδηλατόδρομοι να χρηματοδοτούνται από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Γιατί η Ευρώπη ε, έχει ένα πρόγραμμα με ελέγχου, με γραφειοκρατία και τελικά όλο αυτό το, το σύστημα κοστίζει, έτσι. Αυτό είναι και το πρόβλημα, λέει Το πρόβλημα είναι ότι ένα προπολογισμό, ή μάλλον μια πολιτική, λειτουργεί και με το καρότο και με τον μπαστούνι. Αλλιώ δεν λειτουργεί. Αν υπάρχει μόνο ε, ο βούρδουλα, α πούμε, μόνο οι ρυθμίσει και οι κανόνε, κάποια στιγμή ο κόσμο μπουχτίζει. Στοπ. Θα πρέπει να υπάρχουν και κανόνε, αλλά θα πρέπει να βοηθούμε και τι τοπικές αρχές κτλ. τα λοιπά, χαϊδεύουμε και τα πάντων, αρχίζω να διολυσταίνω λιγάκι και να ξεφεύγω. Τέλο πάντων, αυτή η συζήτηση είναι μεγάλη, αλλά κάπω πρέπει να γίνει. Ε, το θέμα των ποδηλατόδρομων το χρησιμοποίησα μόνο και μόνο για να δούμε ότι η συζήτηση είναι πολύ πιο περίπλοκη από αυτό που φανταζόμασταν στην αρχή. Έτσι, δεν ήθελα, δεν ήθελα να, να μιλήσω, να μπω σε μια πολεμική για τους ποδηλατόδρομους τώρα. Η Κομισιόν σίγουρα για του ποδηλατόδρομους θα κανονίσει ένα ε, μία νομοθεσία για το, την, ε, το πλάτος του ποδηλατόδρομου, ε, για την σύσταση και υφή ας πούμε των υλικών, ε, με έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου, ούτω ώστε... Ε, κοιτάξτε κυρία αυτή, εάν δεν χρηματοδοτήσετε τους ποδηλατόδρομους, η, η Κομισιόν ούτως ή άλλως θα τα καθορίσει όλα αυτά, χωρίς να βάλει και ούτε μία δεκάρα από την τσέπη της. Α, το Κοινοβούλιο όμως θα το επιτρέψει αυτό. Λοιπόν, για να απαντήσω τώρα σε κάποιον άλλον ευρωβουλευτή που έλεγε θα έχουμε τα μέσα ευελιξίας ε, το 1 δισεκατομμύριο ας πούμε για τους Έλληνες που έχουν υποδεχτεί 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Η, Ισπανίδα Ευρωβουλευτής είπε πολύ σωστά ότι θα πρέπει να έχουμε όλη συνείδηση ότι, ότι φτάσαμε στο όριο του προϋπολογισμού που μας επιτρέπει το πουδου που 2014-2020. Είμαστε μόνο στις αρχές του 2016 και έχουμε ακόμα τρεις ε, οικονομικές χρήσεις να ολοκληρώσουμε. Έχουμε χρησιμοποιήσει όλο το περιθώριο ευελιξίας ήδη. Έχουμε ε, χρησιμοποιήσει σχεδόν όλες τις οροφές, όλα τα ανώτατα όρια. Έχουμε εξοδέψει μία σειρά από... Ε, ας πούμε, κονδύλια σε δια... και τα έχουμε βάλει σε διάφορα ταμεία, από εδώ και από εκεί, ας πούμε, για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε λοιπόν ότι είμαστε πολύ κοντά στην απόλυτη δημοσιονομική κρίση. Βεβαίως υπάρχουν πολλές λύσεις οι οποίες υπάρχουν μπροστά μας, θα πρέπει να εγγύψουμε και να τις δούμε, αλλά είναι μόνο η αρχή της συζήτησης. Φυσικά θα ήθελα η συζήτηση αυτή να γίνει με τα εθνικά κοινοβούλια και να σας πω ότι το θέμα των ιδιών πόρων είναι μείζον. Εάν δεν βγούμε από αυτή την κατάσταση, ε, δίνω την επιταγή μου εγώ, ας πούμε, το κράτος μέλος Χ και με αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνουμε το 90% του προπολογισμού, έτσι, μέσω των ιδιών πόρων δηλαδή. Τότε είμαστε σε αένα η κρίση. Υπάρχει αδιαφάνεια, υπάρχει αένα η αναζήτηση ενός νέου, μια νέα ισορροπία στον προπολογισμό και ποτέ θα τη βρίσκουμε. Και φυσικά σύμφωνα με τον Πρόεδρο για τη σημασία του ότι δεν μπορούμε κάθε τόσο να χώνουμε το χέρι, ας πούμε, στη τσέπη των Ευρωπαίων φορολογούμενων και να τους παίρνουμε λεφτά, θα πρέπει να βρούμε λοιπόν μια φορολογία η οποία θα βαραίνει, ας πούμε, τις ε, πολυεθνικές, οι οποίες έχουν κλέψει. Πηδώντας από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, ε, φόρος στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, υπάρχουν και άλλες λύσεις για να βρούμε μια φορολογία που δεν θα βαραίνει μόνο τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Είναι απλή η σύνταγη, λιγότερο από τον ε, φορολογούμενο να ζητήσουμε και περισσότερο από αυτούς που έχουν, από τους έχοντες. Είναι δύσκολα όλα αυτά. Κλείνουμε λοιπόν την πρώτη, το πρώτο τμήμα της συνεδρίασής μας και περνάμε στα πιο συγκεκριμένα θέματα τώρα γιατί τώρα τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσουμε δεν είναι καθόλου απλά. Το θέμα είναι να βρούμε κάποια ισορροπία μεταξύ των νέων κατεπηγών των αναγκών και των κονδυλίων που υπάρχουν μέσα στα πλαίσια του δευτέρου τμήματος του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου του 2014-2020. Το πρώτο τμήμα είναι νέες χρηματοτικές ανάγκες για την αντιμετώπιση των ε, προσφυγικών θεμάτων και η κυρία Ρόιγκ Γκρανζόν από την Υπάτη Αρμοστία για τους πρόσφυγες θα παρουσιάσει το θέμα αυτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων, εκπρόσωπο την είπατε αρμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες. Σας καλημερίζω και σας ευχαριστώ που μου δώσατε την τιμή να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση. Επιπλέον θα ήθελα λόγω της πρόσκλησης αυτής ε, της Επιτροπής Προϋπολογισμού να πω ότι εμείς ε, ε, στα Ηνωμένα Έθνη δεχόμαστε πολύ συχνά πολλές φορές κριτική λόγω των δράσεων του ΟΗΕ και των δράσεων που έχουμε στις διάφορες χώρες. Ε, τώρα, η κρίση που αγγίζει τα τελευταία χρόνια την Ευρώπη, που πλήττει την Ευρώπη και που έχει πολύ σημαντικές διαστάσεις, μας ε, δίνει στην ουσία τη δυνατότητα να στραφούμε προς τον ΟΗΕ, μια δομή που έχει την ε, επιχειρησιακή και λειτουργική δομή να μας βοηθήσει να υποστηρίξουμε τους εκτοπισμένους. Τα τελευταία χρόνια, από το καλοκαίρι του 2015, ε, ουσιαστικά με μεγαλύτερη ένταση, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με μία μεγαλύτερη ανάγκη λόγω της ε, κρίσης αυτής που έχει ε, διαστάσεις που δεν είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν. Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι δήμοι, στην ουσία έρχονται αντιμέτωποι με μια πολύ μεγάλη πίεση, όπως και η κοινωνία των πολιτών, που δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Η πανεπιστημιακή και όλος ο κύκλος των ακαδημαϊκών συμφωνούν πως αν δεν ε, επενδύσουμε σε ένα θεωρητικό πλαίσιο ε, έτσι ώστε να υπάρξει μια καινοτομία ε, και καλύτερες λύσεις για το προσφυγικό και το, την εκτόπιση των πληθυσμών θα έχουμε διαδοχικές τέτοιες κρίσεις. Τώρα αυτή η συζήτηση για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ένα θέμα επί το οποίο εργαστήκαμε από κοινού, ουσιαστικά για τα εσωτερικά κονδύλια, ε, τα κονδύλια δηλαδή της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις που έχουν και παγκόσμιο επίπεδο. Ε, ε, είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε πολλές αναθεωρήσεις του προπολογισμού και δεν είναι τώρα αυτή η ευκαιρία μόνο μία ευκαιρία για να κάνουμε έναν απολογισμό, αλλά είναι και μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να θέσουμε προτεραιότητες και να δούμε πώς θα γίνει στο μέλλον ε, ο προϋπολογισμός και ο κύκλος του έτσι ώστε να αντιμετωπίζει τις πραγματικές ανάγκες. Να μπορούμε να προβλέπουμε. Είδαμε λοιπόν ότι τα μέσα ευελιξίας χρησιμοποιήθηκαν πλήρως, οπότε τώρα ίσως θα πρέπει να δούμε κάπως διαφορετικά τα πράγματα και να εισαγάγουμε νέους μηχανισμούς. Επίσης θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ε, την εξής πληροφορία. Η έναρξη του νέου κύκλου το 2014 ήταν δύσκολη, ειδικά για τους νέους τίτλους ε, άσυλο, μετανάστευση, ενσωμάτωση. Ε, είναι θέματα της ε, Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων χρειάστηκε μία αναδιάρθρωση που οδήγησε τα κράτη-μέλη στο να χρησιμοποιήσουν ένα νέο τρόπο λειτουργίας. Το θέμα αυτό ήδη συζητήθηκε, δηλαδή τα 24 δις που έχουν μείνει απλήρωτα για το 2014 και μιλήσαμε και γι' αυτό το χάσμα μεταξύ της δυνατότητας πληρωμών και των δεσμεύσεων που έχουν αναλυφθεί. Όλα αυτά είχαν πολύ σημαντικές επιπτώσεις ε, για τους ανθρωπιστικούς οργανισμούς ε, και όλες αυτές τις δράσεις τις οποίες συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε έλλειψη μέσων ε, στο πεδίο. Αυτό είχε άμεση επίπτωση λοιπόν στην τρέχουσα κατάσταση. Για να είναι σωστά διαρθρωμένη η συζήτηση θα πρέπει να διαχωρίσουμε τις κρίσεις αυτή που έχει να κάνει με το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τη διαχωρίσουμε από αυτή που υπάρχει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεταναστευτική κρίση που πλήττει την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, το γεγονός ότι φτάνουν τόσοι πρόσφυγες στα σύνορα της Ευρώπης, ε, πρέπει να το διαχωρίσουμε από τις κρίσεις στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή, όπου οι προκλήσεις είναι τελείως διαφορετικές. Ας ξεκινήσω λοιπόν με την κρίση ε, στην Ευρώπη και θα σας δώσω και κάποια νούμερα. Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν φτάσει από το καλοκαίρι ή λίγο πριν το καλοκαίρι και ως το τέλος του έτους στην Ευρώπη έφτασαν με για να είμαι πιο συγκεκριμένη. Ε, ακόμα περισσότεροι ήρθαν ε, από τα χερσαία σύνορα. Υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα και 82.000 άτομα έχουν έρθει μέσω της Ελλάδος και της Ιταλίας, οι περισσότεροι από την Ελλάδα. Το 80% αυτών των αριθμών στην ουσία αφορούν ανθρώπους που προέρχονται από τις 10 πιο παραγωγικές χώρες σε επίπεδο προσφύγων, χώρες προέλευσης. Άρα είναι κυρίως κρίση προσφυγική και όχι μεταναστευτική. Να σας ε, θέσω και κάποια ερωτήματα και όχι τόσο συστάσεις ε, για να τα σκεφτούμε περισσότερο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε ε, έκτακτα μέτρα και να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση ως έκτακτη ή θα πρέπει να έχουμε μια πιο διαρθρωμένη προσέγγιση στο μέλλον δεν ελπίζουμε ότι η κρίση θα συνεχίσει σε καμία περίπτωση. Απλώς ε, ο αριθμός των ανθρώπων που πρόκειται να έρθουν ε, στο μέλλον, ε, πολύ φοβόμαστε ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερος σύμφωνα με τις αναλύσεις. Δεύτερον, και αυτό είναι ένα θέμα που έθιξαν και στα συμπεράσματά τους οι προηγούμενοι ομιλητές. Αυτό το αυτός ο μηχανισμός ε, θα πρέπει να είναι εθνικός, ευρωπαϊκός ή θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός. Και το θέμα της προστιθέμενης αξίας. Εφόσον υπάρχουν τόσοι ε, βουλευτές εδώ από τα Εθνικά Κοινοβούλιο, είναι πολύ σημαντικό να θέσουμε αυτό το ερώτημα. Είναι προφανές ότι ο στόχος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ούτε ήταν ποτέ ούτε θα πρέπει να είναι να γίνει υποκατάστατο των εθνικών προϋπολογισμών που υπάρχουν ήδη για να αντιμετωπιστούν τέτοιες καταστάσεις. Όχι βέβαια όταν είμαστε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κρίσης, αλλά σε κάθε περίπτωση ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν πρέπει να είναι υποκατάστατο υποκατάστατο των εθνικών προϋπολογισμών. Θα πρέπει να είναι μια προστιθέμενη αξία. Αν μου επιτρέπετε, συμπληρωματικά υπάρχουν δύο τρόποι να προχωρήσουμε. Είτε από τον, ε, προέρχομαστε από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό είτε από τα κράτη-μέλη, όπως είδαμε και αυτά που έγιναν την περασμένη εβδομάδα στην Τουρκία. Υπάρχει στην Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Ο συντονισμός λοιπόν ήταν ε, αυτό ε, που προκρίθηκε και από εκεί προήρθε το Trust Fund φαντάζομαι. Ναι, το Trust Fund στην ουσία ήταν ένας τρόπος για να έχουμε ένα προσάρτημα ας πούμε στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αναλύσουμε τα κονδύλια. Ναι, και να τα συντονίσουμε, ναι, ε, για να υπάρχει καλύτερο συντονισμός. Ναι, να τα έχουμε όλα συνδυασμένα. Ναι, δεν μίλησα για Trust Fund, αλλά είναι και ένας από τους στόχους, ίσως και μια πρόκληση για μια κρίση που είναι ε, κοντά στην Ευρώπη αλλά και για τις πιο μακρινές κρίσεις. είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ο 21ος δωρητής πέρα των υφιστάμενων 28. Τίθεται λοιπόν αυτό το ερώτημα. για την εσωτερική κρίση τώρα της Ευρώπης, αλλά ένα ενδιαφέρον ερώτημα είναι εάν θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα μέσονος μηχανισμός επέμβασης για την ανθρωπιστική βοήθεια. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε ε, εσωτερικό επίπεδο στην κοινότητα, αλλά αν η κατάσταση ας πούμε στην Ελλάδα ε, επιδεινωθεί λόγω κλεισίματος των ε, Βαλκανικών συνόρων ή ενός άλλου σεναρίου που δεν ελπίζουμε, θα υπάρχουν άνθρωποι και η Ένωση θα είναι μπλοκαρισμένη σε αυτόν τον μηχανισμό της έκτακτης ανάγκης. Έτσι λοιπόν, μέσα από την ευελιξία, ίσως θα πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία η οποία δεν θα είναι ποτέ ε, στο επίπεδο να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Τώρα για την εσωτερική κρίση, άλλη μια παρατήρηση. Όλο και περισσότερο διαβάζω ε, την έκκληση προς τους πιστοτικούς οργανισμούς, ε, μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και αναρωτιέμαι πώς μπορεί αυτό να διαρθρωθεί και να συνδυαστεί. Όπως σας είπα και πριν λέει ο Πρόεδρος, για να κερδίσουμε χρόνο, έχουν την εμπειρογνωμοσύνη που θα μας επέτρεπε να πάμε πιο γρήγορα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό σε αντίθεση με στην ουσία με την κατάσταση που υπάρχει λόγω της σχέσης μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία μας ε, επιτρέπει, δεν μας επιτρέπει να έχουμε μια σωστή αντιμετώπιση. Χρειαζόμαστε λοιπόν την εμπειρογνωμοσύνη αυτών των οργανισμών για να έχουμε πιο γρήγορες ε, πολιτικές αποφάσεις. Σε ποιο θέμα εμπειρογνωμοσύνη. Για τα σχολεία, ας πούμε. Στην Τουρκία υπάρχουν 15.000 παιδιά που δεν πάνε στο σχολείο και αυτά μπορεί να είναι μια γενιά χαμένη στο τέλος. Ναι, συμφωνώ. Εντάξει, είναι άλλο ένα στοιχείο που μπαίνει στη συζήτηση και σε αυτή την πολύπλοκη κατάσταση. Έχω ήδη μιλήσει 11 λεπτά και γι' αυτό θα μιλήσω τώρα για τις κρίσεις στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέθηκε το θέμα του Trust Fund. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ λίγη χρηματοδότηση από την πλευρά των κρατών μελών. Είναι ένα trust fund το οποίο είναι εσωτερικό ε, είναι διάφορα ε, κονδύλια που προέρχονται από τους διάφορους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα δεν είναι να δημιουργήσουμε το Trust Fund, είναι να του δώσουμε ε, τη χρηματοδότηση που χρειάζεται, τα κονδύλια που χρειάζεται. Ναι, ακριβώς, γιατί υπάρχει και αυτό το φαινόμενο της χιονοστιβάδας που προκαλείται. Και δεν συμβαίνει αυτό αυτή τη στιγμή. Ωραία, επιτρέψτε μου να κάνουμε τελευταία παρατήρηση Όπω είπε και ο προηγούμενο επίτροπο, ο κύριο Κουτιέρε, ο οποίο ε, είχε μιλήσει στο Διεθνέ Οικονομικό Φόρουμ πέρυσι, νομίζω, στον ταβό, που είχε να κάνει με τη νέα αρχιτεκτονική της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής βοήθειας ε, που είχε να κάνει και με αυτή την σύνοδο κορυφής για την ανθρωπιστική κρίση στην Κωνσταντινούπολη τον Μάιο. Βρισκόμαστε λοιπόν σύμφωνα με αυτό σε μια κατάσταση που η, ζήτηση ας πούμε είναι πολύ μεγαλύτερη από την πρόσφορα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε αυτές τις εκκλήσεις μεταξύ των οργανισμών στα Ηνωμένα Έθνη για την αντιμετώπιση κρίσεων. 50, ε, ε, στο 50-60% των περιπτώσεων ακόμα και στα 2 τρίτα. Υπάρχει υποχρηματοδότηση, υπο-υποχρήματοδότηση, άρα πρέπει να σκεφτούμε ξανά την αρχιτεκτονική της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού. Σύμφωνα με την παραδοσιακή προσέγγιση υπάρχουν οι φορολογούμενοι τους οποίους αναφέραμε και πριν, υπάρχουν και οι ανθρωπιστικοί κοινωνικές οργανώσεις, κυβερνητικές και μη κυβερνητικές και υπάρχουν και οι πληθυσμοί των χωρών υποδοχής που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος, αλλά και οι δωρητές που προσπαθούν να συντονίσουν όλα αυτά. Όλα αυτά τα υποστηρίζουν οι φόροι, οι φορολογούμενοι. Άμεσα των Ευρωπαίων, αν μιλάμε για την Ευρώπη. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα αυτού του φόρουμ, είναι απαραίτητο να επανεξετάσουμε αυτή την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και να συμπεριλάβουμε και τον ιδιωτικό τομέα ως ένα νέο παράγοντα, ένα νέο παίκτη. Ο ιδιωτικός τομέας στην ουσία δεν είναι αυτός που κακώς νοούμε πολλές φορές ως μια ξεχωριστή οντότητα, είναι οι πιο ισχυροί αυτού του πλανήτη που θέλουν να εμπλακούν. Και σας διαβάζω ε, το τέλος. Ο Bill Gates ας πούμε ναι, και αυτός, ε, ο οποίος λέει και το λέει στα αγγλικά, αν μου επιτρέπετε, ότι με τους φόρους που πληρώνουν στην Ευρώπη μπορούμε και εμείς να συμμετέχουμε. Κοιτάξτε, ε, σε ένα κόσμο που η τελευταία εφαρμογή κινητών ε, μπορεί να φέρει δισεκατομμύρια δολάρια, μπορούμε να δώσουμε κάποια χρήματα για τους χώρες που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε τους πόρους και την τεχνογνωσία ως παγκόσμια κοινωνία και να κάνουμε μια τεράστια διαφορά στο επίπεδο διαβίωσης των προσφύγων. Αυτό δεν θα γίνει μέχρι ο ιδιωτικός τομέας να αποφασίσει ότι πρέπει να συμμετάσχει και να γίνει η κινητήρια δύναμη σε αυτή τη δυνατό, την ε, προσπάθεια αντιμετώπισης. Φαίνεται λοιπόν ότι από τη Συρία καταλάβαμε πως ε, η προσέγγιση που υπάρχει ως τώρα δεν λειτουργεί. Καιρός να βρούμε μια καινούρια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και ο δεύτερος ομιλητής μας που εκπροσωπεί τις ε, είναι Γενικός Γραμματέας Συμβουλίου των, Εθνικών, των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιοφών ο κύριος Βαλιέ. Ζήτησε η προηγούμενη ομιλήτρια να κάνουμε κάποια βελτιστοποίηση, λέει, παρεμβαίνει ο πρόεδρος. Και όχι καταναγή μόνο χορηγίες. Οι Ευρωπαίοι μπορούν να δώσουν τα καλά εργαλεία σε όλους τους εμπειρογνώμονες βελτιστοποίηση να το κάνουν. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να γίνει καλύτερη βελτιστοποίηση, λέει ο πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, Ευρωπαίοι και Εθνικοί Κοινοβουλευτικοί, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την ε, πρόσκληση που με απευθύνατε και ιδιαίτερα την κυρία Τομά και τον κύριο Όλμπριθ για την πρόσκληση αυτή στην ε, συνεδρίαση αυτή που αφορά και τις δράσεις των Δήμων και Περιφερειών σε σχέση με την αντιμετώπιση της έκτακτης ανθρωπιστικής κρίσης λόγω του προσφυγικού ρεύματος. Το Συμβούλιο των Κοινοτήτων και Περιφερειών της Ευρώπης, από το οποίο είμαι Γενικός γραμματέα, εκπροσωπεί 55 ευρωπαϊκές εθνικές ενώσεις, δήμων, πόλεων και περιφερειών σε 41 χώρες, μεταξύ των οποίων και 48 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επίση και χωρών των Βαλκανών, νέων της Τουρκίας και την Ουκρανία. Έχουμε έτσι μια κοινότητα 150.000 τοπικών αρχών στην Ευρώπη, που καλύπτει το σύνολο της ε, Ευρώπης. Ενώπιον της κρίσης αυτής, όπως ενώπιον οποιασδήποτε σοβαρής κρίσης, οι τοπικοί εκλεγμένοι έχουν δείξει μεγαλύτερη ευαισθησία από ότι οι ομόλογοι του σε επίπεδο Εθνικού Κοινοβουλίου, εθνικού, Εθνικών Κυβερνήσεων βέβαια, ή εγκύτητα το, απαιτεί, το απαιτεί αυτό. Η ανάγκη για πόρους είναι ένα πραγματικό ερώτημα. Και εδώ πραγματικά εμπλέκεται και η ίδια ιδέα του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Γι' αυτό μέσα στα πλαίσια του πακέτου για την καλύτερη διαχείριση τη μετανάστευση που θα ξεκινήσει το Μάρτιο ή τον Απρίλιο, οι τοπικέ αρχέ θέλουν να αγωνιστούν μαζί με το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η κρίση των μεταναστών και συγχρόνω να γίνει η, η απαραίτητη μεταρρύθμιση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου του επόμενου μήνε. Πέραν αυτού, από την έναρξη της κρίσης το, το, την άνοιξη του 2015 έχουμε δημιουργήσει εργαλεία αξιολόγησης <clears throat> επιτόπιας και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε βοήθεια στους λήπτες αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται από το τοπικό επίπεδο. Για να συμπληρώσουμε αυτήν τη συλλογή στοιχείων θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο το οποίο να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες και επίσης να βοηθήσει τους κλίμους και τις κοινότητες για να υπάρχει η βελτίωση των πρακτικών σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση των των άσυλων. <clears throat> Με την κρίση των ε, προσφύγων, το δημοσιονομικό πλαίσιο έχει φτάσει στα όρια του. Από τον Ιανουάριο του 2015 έχουμε πάνω από 710.000 ετούντες άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στα ανατολικά είτε στα νότια σύνορά της. Από το 2017, αν δεν υπάρξει καμιά λύση, θα φτάσουν σε περίπου 3 εκατομμύρια που προερχόνται από ζώνες πολεμικές και θα είναι στα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η κρίση προστίθεται στην χρηματοοικονομική κρίση, αλλά συμφωνούμε με την ανάλυση του Πρόεδρου Γιούνκερ, ο οποίο αναγνώρισε όταν μιλούσε ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι τα, εξαιρετικέ συνθήκε απαιτούν εξαιρετικά μέτρα. Πράγματι, οι πόροι που είναι διαθέσιμοι στο τωρινό δημοσιονομικό πλαίσιο, ακόμα και αν χρησιμοποιηθούν απόλυτα όλα τα περιθώρια τα οποία υπάρχουν για την ευελιξία, θα φανούν μάλλον ανεπαρκή τα επόμενα χρόνια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό οι δήμοι οι οποίοι συμμετέχουν στα προγράμματα επανεγκατάστασης ή τα συστήματα ποσοστώσεων για του πρόσφυγε, αντιμετωπίζουν πολλά απρόβλεπτα ε, έξοδα τα οποία δεν καλύπτονται πλήρω ούτε από τις κεντρικές κυβερνήσει ούτε από κανέναν άλλο. Δεν υπάρχει περιπτώσει, κάποια κάλυψη από τις εθνικέ αρχέ. Ενώ σε πολλέ χώρε τα χρήματα τα οποία δίδονται από τι προς τις ε, τοπικές αρχές για κοινωνικές παροχές έχουν μειώσει, αυτές οι χώρε βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ε, υποδοχής των προσφύγων. Πρόκειται για την Ελλάδα, αλλά και για τη Φιλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία. Και εκεί είναι φανερό ότι τα έσοδα των τοπικών αρχών καταραίουν αυτή τη στιγμή. Και επίση, βάσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, οι τοπικέ αρχέ θα πρέπει να προστατεύσουν του ασυνόδευτου ανήλικου, κάτι το οποίο σημαίνει μια υπερβολική, ε, ένα υπερβολικό οικονομικό βάρος εάν δεν υπάρξει καμία βοήθεια από τις εθνικές κυβερνήσεις. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να γίνει να αναγνωριστεί. Είναι σαφέ ότι το συνολικό πλαίσιο το οποίο έχει συμφωνιστεί για το διάστημα 2014-2020 είναι ανεπαρκέ για να μπορέσει να αντιμετωπίσει πολλαπλέ κρίσει τι οποίε αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τοπικέ αρχέ δεν έχουν του απαραίτητου πόρου είτε ω χώρε πρώτη άφηξη, χώρε διέλευση ή χώρε τελικού προορισμού δεν υπάρχει χρηματοδότηση σε τοπικό επίπεδο για να μπορέσει να δοθεί η βασική βοήθεια στους πρόσφυγες, δεν υπάρχουν στέγα, ε, καταλήματα, στέγαση, ψυχολόγοι, ε, διδάσκαλοι, κοινωνική ε, λειτουργή και διερμηνής. Για παράδειγμα, η περίπτωση τη Γερμανία που είναι η χώρα η οποία έχει υποδεχθεί το μεγαλύτερο μέρο των προσφύγων. Η κατανομή του κόστου μεταξύ των διαφόρων επίπεδων ευθύνη είναι ω εξή. 15 δισεκατομμύρια έχει κοστίσει στην Γερμανία, από τα οποία το 2015 10 δισεκατομμύρια από τις τοπικές αρχές και 5 από τα Λέντερ και το ομοσπονδιακό επίπεδο. Για τους πρόσφυγες του 2016 το κόστος μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 9 και 25 δισεκατομμυρίων ευρώ και το μεγαλύτερο από μέρος από αυτά πρέπει να καλυφθεί από το τοπικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι αν λάβουμε υπόψη το συνολικό αριθμό των προσφύγων που έχουν φτάσει το 2015 μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσθεθεί να προσταθούν 30 δισεκατομμύρια ευρώ στον προπολογισμό τη για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει πλήρω την κρίση. Υποστηρίζουμε λοιπόν αυτά που λένε οι συγητέ, ότι πρέπει να υπάρξουν πρόσθετε και έκτακτε πηγέ χρηματοδότηση. Επιπλέον, πλέον τη ευελιξία είναι απαραίτητο για να μπορέσουν να υλοποιηθούν αυτέ τι πολιτικέ να υπάρχει και η καλύτερη χρηματοδότηση των αναγκών των τοπικών αρχών. <clears throat> Θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε να εξετάσουμε έκτακτα μέτρα για να αυξηθούν οι ήδη πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης να βελτιωθεί η χρήση άλλων ε, υπαρχουσών πηγών εσόδων και να εξετάσουμε δυνατότητα αύξηση φορολογία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ζητούμε από την ομάδα υψηλού επίπεδου για του ίδιου πόρου να επιταχύνει τι εργασίε τη και από το Συμβούλιο να δείξει φιλοδοξίε στι επόμενε συνεδριά του. Υποστηρίζουμε μία ε, χρηματοδότηση από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είτε <clears throat> με ένα ειδικό ευρωπαϊκό δάνειο είτε με ένα προσωρινό φόρο για την ενέργεια επί τη βάση της ε, περιεκτικότητας σε άνθρακα βασιζόμενοι στη χαμηλή τιμή του πετρελαίου αυτή τη στιγμή. Επίσης θέλουμε τα κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν στου μηχανισμού επανεκατάστασης να ωφεληθούν από αυτή την αύξηση των πόρων με την προπόθεση να υπάρξει σωστή κλίδα κατανομή μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δώσει δάνεια σε μηδενικό επιτόκιο για να μπορέσουν να υπάρξουν περισσότερα καταλήμματα, ένα τμήμα των οποίων μπορεί να δοθεί στου πρόσφυγε. Μέσα στα πλαίσια του τωρινού συστήματο χρηματοδότηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει κανένα ειδικό πόρο ο οποίο έχει τεθεί κατά μέρο για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Γι' αυτό ζητούμε από το Κοινοβούλιο, από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο με την υποστήριξη πιστεύω των Εθνικών Κοινοβουλίων στη διαδικασία μεταρρύθμιση <clears throat> του δημοσιονομικού πλαισίου πέραν των μέτρων εκτάκτη ανάγκη για ε, την εγκατάσταση των προσφύγων να υπάρξουν και περαιτέρω πόροι για την ενσωμάτωσή του σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Επίση, οι πόροι οι οποίοι έχουν υποχρησιμοποιηθεί θα πρέπει να ανακατευθυνθούν και να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ να αντιμετωπίσουν καλύτερα τι ευθύνε του στον τομέα αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια σειρά από προτάσεις για καινοτομίε στον αστικό χώρο που να υλοποιηθούν από το ΦΕΝΤΕΡ για να υπάρξει η δυνατότητα στις πόλεις και στις κοινότητες να δώσουν καταλήμματα στους ε, πρόσφυγες και χρειάζεται να πάρουμε και διαφορετικό χαρακτήρα όλα αυτά. Επίση υπάρχει και ένα περιθώριο δράση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε συνέργειε μεταξύ των μηχανισμών χρηματοδότηση που υπάρχουν όπω είναι το Ταμείο για την Εσωτερική Ασφάλεια, το ΑΜΥΦ, το οποίο είναι το Ταμείο για το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ολοκλήρωση, το Κοινωνικό Ταμείο και το Περιφερειακό Ταμείο. Θέλουμε να ενισχύσουμε την αρχή τη επικουρικότητα και τη εταιρική σχέση ώστε να υπάρξει μια καλύτερη προσέγγιση σε πολυεπίπεδο σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνηση που υπερλαμβάνει και τι αποφάσει για τον προπολογισμό και του πρόσφυγε. Αυτή η, η προσέγγιση θα πρέπει να καλύψει όχι μόνο την εγκατάστασή του, αλλά και τα άλλα μέτρα σε εθνικό επίπεδο, αλλά επίση όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των μηχανισμών χρηματοδότηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητάμε να υπάρξει ευελιξία σε ό,τι αφορά το, το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη για του ε, Δήμου που αντιμετωπίζουν μεγάλο αριθμό προσφύγων και έχουν έλλειψη πόρο Θεωρούμε ότι η συνεργασία μεταξύ των πόλεων υποδοχής και των πόλεων προέλευσης μπορούν να συμβάλλουν ιδιαίτερα να συμβάλλουν στην ενσωμάτωση των ε, προσφύγων και την επιστροφή τους όταν τελειώσει η κρίση. Επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει αυτούς τους δεσμούς, να τους ενισχύσει και να δημιουργήσει και πρωτοβουλίες καλύτερης ε, συνειδητοποίησης όπως το πρόγραμμα DEAR για τα προγράμματα ανάπτυξης. Και εν τέλει, για κλείνοντα θέλω για μια ακόμα φορά να υπογραμμίσω το ρόλο των δημάρχων και των τοπικών εκλεγμένων, των τοπικών και εδαφικών αρχών, που πολλέ φορέ αντιμετωπίζουν αφόρητε ανθρωπιστικέ κρίσει, αλλά που αντιμετωπίζουν τις και αυτό με του Δημάρχου τη Λέσβου, τη Κόρτη, τη Ναθηνών, τη Λαμπεδούσα, του Καλέ, για να σα δώσω μόνο μερικά παραδείγματα. Είμαστε υπερήφανοι για τον αγώνα τους υπέρ των αξιών που έχουν οικοδομήσει στην Ευρώπη μα και το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης είναι στο πλευρό τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν να δίνουν το μήνυμα ανθρωπιστικό, ανθρωπιστικό μήνυμα υπέρ του ευρωπαϊκού εγχειρήματο και σας ευχαριστώ για την προσοχή. Euh, για αυτές τις διαφορετικές παρατηρήσεις. Εσείς μια και είσαστε όλοι μέλη κοινοβουλευτικών επιτροπών προϋπολογισμού, έχετε κάνει, ξέρετε από δύσκολε ε, επιλογές στην πολιτική. Και εδώ και ένα χρόνο αντιμετωπίζετε αλλεπάλληλες απογοητεύσεις. Αλλά θα πρέπει να κάνετε έτσι, επιλογές και με τα μέσα που διαθέτουμε να επιλέξετε. Θα ήθελα όλοι τώρα να κάνετε τις παρεμβάσεις σας το πολύ μέσα σε δύο λεφτά, αν μπορείτε βέβαια, γιατί έχουμε καθυστερήσει. Πρώτος, ο μιλητής και ο Μυρόσκαβα Νάγκελ. Ζητώ συγγνώμη που σας το σκότωσα το όνομα. Είναι Πολωνός Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μέλος του ΕΛΚΑ. Η κυρία. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Ο σκοπό του κοινοτικού προπολογισμού είναι να μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε τι προτεραιότητε τη Ένωση Στο όνομα όλων των Ευρωπαίων πολιτών και για όλου του Ευρωπαίου πολίτε. Γι' αυτό οι δαπάνε υπό τον προπολογισμό θα πρέπει να υπόκεινται σε δημοκρατικό έλεγχο. Και επίση θα πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση ε, για το κατά πόσον ε, εκπληρώνονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η πολιτική συνοχής έχει αποδείξει την αξία της ω τμήμα της διαδικασίας ένταξης. Η αξία της λοιπόν είναι τεράστια, γιατί φαίνεται ε, με γυμνό μάτι και τη βλέπουν οι πολίτες. Αλλά υπάρχει ένα ναι μεν αλλά. Για προγράμματα του ορίζοντα 2014-2020 που δεν έχουν ακόμα πλήρως υλοποιηθεί, υπάρχει ανάγκη να ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα για τομείς όπως ε, η κρίση της μετα μεταναστευτική κρίση. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν τα κονδύλια για να τα ξοδέψουμε εκεί στι νέε προκλήσει γιατί είναι αυτό το θέμα θέμα αξιοπιστίας τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αξιοπιστία σημαίνει ε, ναι, να αντιμετωπίσει τι νέε ανάγκες, αλλά και να, να συνεχίσει τι δεσμές που έχει αναλάβει και να τι σεβαστεί, κύριε Λεβαντόφσκι. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Έχω μία ερώτηση τώρα. Πώ βλέπετε εσείς κυρίε και κύριοι τη δυνατότητα δαπανών ε, για νέα θέματα, για νέους τομείς, χωρίς να κλέψουμε, αν θέλετε, να πάρουμε λεφτά από τα υπάρχοντα ταμεία. Χωρίς βεβαίως να θέσουμε να αμφιβόλω την, ε, την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας. Την ΚΕΠΑ δηλαδή. Ευχαριστώ. Ολαβία Λανίσιλα μέλος ε, του Φιλανδικού Κοινοβουλίου, Επιτροπή Οικονομικών, Δημοσιονομικών. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε. Σύντομα. Μία γενική αρχή. Χρησιμοποιούμε δημόσιο χρήμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να, να υπάρχει και κανονικότητα, τακτικότητα και διαφάνεια και λογοδοσία. Αυτά θα πρέπει να υπάρχουν. Είναι εκ των όνου κάνευ. Για τη μεταναστευτική κρίση και τη χρήση των ε, δημοσίων κονδυλίων για την υποδοχή των ε, προσφύγων, αυτή είναι τεράστια πρόκληση. Γιατί θα πρέπει να ληφθούν πολύ γρήγορα αποφάσεις, ε, καινοτόμες αποφάσεις, αποφάσεις που δεν έχουμε ξαναπάρει ποτέ και αναπάντεχες. Ε, είναι πρόβλημα εθνικό και ευρωπαϊκό και επομένως αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, από τον κοινοτικό προπολογισμό. Επίσης, σε εθνικό επίπεδο διερωτώμεθα πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τι δαπάνε όταν υπολογίζουμε τα δημοσιονομικά ελλείμματα, ας πούμε, ή τα κριτήρια τα οποία θα εφαρμόσουμε, τα κριτήρια του Άμστερνταμ, ας πούμε, για τον προϋπολογισμό. Εκεί χρειαζόμαστε συντονισμό. Και είναι κλασικό αυτό το θέμα, το οποίο εξετάζουν ας πούμε, τα, και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τις ε, κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ένωσης και τις αποφάσεις που λαμβάνει το Συμβούλιο. Και το βασικό ερώτημα είναι πολύ σωστό. Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε νέους τρόπους χρηματοδότησης, νέα εργαλεία. Μια άλλη ερώτηση, στα πλαίσια των δαπανών αυτών, ποια είναι η επίπτωση που έχουν αυτές οι δημόσιες δαπάνες. Πρέπει να διαρωτηθούμε τι επίπτωση έχουν αυτές οι δαπάνες. Ο κύριος Μπέγκε έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις συμβολές σας και πολύ σωστά μας υπέδειξε τα προβλήματα η εκπρόσωπος της υπάτησα αρμοστίας. Εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ καμία συνδιάσκεψη που έχω παρακολουθήσει για τα θέματα αυτά του προπολογισμού και ε, συνεδριάσεις χορηγών που άλλα υπόσχονται και στη συνέχεια η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Νομίζω ότι όπως λέτε και εσείς έχουμε κατανοήσει όλοι ότι η διευθυντική κοινότητα τα τελευταία χρόνια έχει πραγματικά με τρόπο ουσιαστικά εγκληματικό έχει παραμελήσει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα όπως με το παγκόσμιο πρόγραμμα τροφίμων. Δεν μπόρεσε λοιπόν να καλύψει τις ανάγκες με τα προ... προβλήματα τα οποία βλέπουμε σήμερα. Έχουμε λοιπόν και το ερώτημα το πολιτικό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε πρώτα απ' όλα. Φτάνουν οι υποσχέσεις οι οποίες έγιναν στη Σύνοδο των Χορηγών του Λονδίνου και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε ενώπιο μας υποσχέσεις οι οποίες είναι αξιόπιστες. Έχουμε εκεί πέρα μια τεράστια ανισομέρεια μεταξύ κρατών μελών από το Λονδίνο που έχουν ε, κάνει μεγάλες υποσχέσεις και άλλες χώρες από την περιοχή της Μέσης Ανατολής που έχουν αγνοήσει τελείως την ανάγκη υποσχέσεων και κονδυλίων. Μήπως πρέπει να έχουμε και ένα μηχανισμό που θα λειτουργήσει καλύτερα και να μην περιμένουμε μήνες για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία της ε, παροχή κονδυλίων και προηγουμένω των υποσχέσεων του. Επίση, το καταπίστευμα για την ε, Αφρική καλύπτει 1,8 δισεκατομμύρια, αλλά προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Και οι εθνικέ συνεισφορέ μέχρι τώρα είναι 81 εκατομμύρια από 1,8 δισεκατομμύρια και έχουμε 16 εκατομμύρια επίσης από, το, από τα, από τα κράτη-μέλη για τα προγράμματα αυτά. Έχουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό ρεύμα, ένα σταθερό ρεύμα από το Ιράκ και μια αύξηση ε, στους πρόσφυγες που έρχονται από τις αφρικανικές χώρες. Και έχουμε να αντιμετωπίσουμε χώρες οι οποίες έχουν αποτύχει ουσιαστικά λίγο πολύ. Με ποιο τρόπο λοιπόν μπορούμε να σκεφτόμαστε για επαναφορά ε, προσφύγων οι οποίοι δεν έχουν καμιά δυνατότητα να ζήσουν, να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν αυτοί συγχρόνως δεν είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε σε βοήθεια οικονομική όπως κάνουμε στην περίπτωση της Τουρκίας και δεν πρόκειται μονάχα για θέματα χρημάτων. Δεν είναι μονάχα χρήματα, είναι, είναι και η σταθερή μας προσέγγιση και οι πιο στενές σχέσεις με γειτονικέ χώρες. Το πραγματικό ερώτημα βέβαια είναι που έχουμε κάνει λάθος σε σχέση με τα σημεία έμφασης της ε, πολιτικής γειτονία μας, η οποία δεν έχει λειτουργήσει. Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε χρηματοδότηση σχεδίων, τα οποία να είναι πιο κοντά στους ανθρώπους επιτοπίως, ή ουσιαστικά θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε σχέδια τα οποία εξυπηρετούν μοναχά τι ολιγαρχίε. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και επίσης πρέπει να σκεφτούμε για την, τον ορισμό των ασφαλών χωρών. Αυτό είναι ένα σίγουρο θέμα, ένα σημαντικό θέμα, αλλά μπορούν ακόμα και οι χώρε που θεωρούμε ασφαλεί, παραδείγματο χάρη στα Βαλκάνια, και αυτέ να βρεθούν σε μια ολιστηρή κατοφέρεια. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε και ποιε είναι οι συνέπειε για το προπολογισμό. Το άρθρο 80 τη συνθήκη Λισαβόνα μιλάει για μια αλληλεγγύη των κρατών μελών μεταξύ του σε περίπτωση μια κρίση ε, προσφύγων. Μιλάει για μια ορθή κατανομή. Και η Κομισιόν είπε ότι και το Περιφερειακό Ταμείο και το Ταμείο Ανάπτυξη μάλλον και τα κονδύλια συνοχή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αντιμετώπιση νέων κρίσεων, όπω η προσφυγική κρίση. Πιστεύω ότι ακόμα και τα διαφορετικά ταμεία, και έρχομαι σε αυτό που είπε ο Πολωνό συνάδελφο, και τα διαφορετικά ταμεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να υπάρξει συγχρηματοδότηση όλων αυτών των ε, θεμάτων. Όταν έχουμε τώρα πρόβλημα με τι ποσοστώσει, Εμείς ξέρουμε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το θέμα ως απλώς μια χαλαρή συνομοσπονδία, ε, μια λέσχη κρατών που θα είναι ανεξάρτητα και όχι σαν μια ενωμένη ομάδα κρατών για να αντιμετωπίσουμε την, ε, την πρόκληση του Πούτιν ή του Τραμπ. Αυτή τη στιγμή η χρηματοδότηση που χρειάζεται για τους πρόσφυγες, όπως είπατε, είναι 30%. Αυτό είναι 1,2 του είναι λιγότερο από 1% του ΑΕΠ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει όμως να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα χρηματοδοτηθούν οι δυνάμεις όπως η Frontex που ελέγχουν τα σύνορά μας και να βοηθήσουμε τις χώρες οι οποίες υφίστανται ένα δυσανάλογο βάρος από το προσφυγικό ρεύμα με ένα ταμείο το οποίο θα είναι ευρωπαϊκό και αλληλεγγύη. Αυτό θα είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Ευχαριστώ. Πώς θα εξασφαλίσουμε εκ νέου την ειρήνη. Γιατί στη Συρία υπάρχουν 8 με 10 εκατομμύρια εκτοπισμένοι. Πολλοί από αυτού ε, συσσωρεύονται στα τουρκικά σύνορα, τα οποία όμω δεν μπορούν να περάσουν πια. <laughs> Νομίζω ότι ο ΙΕ δημιουργεί στρατόπεδα από την πλευρά της ε, Συρίας κοντά στην Τουρκία. Ασχολείται η Τουρκία με αυτό το θέμα. Μάλιστα. Α, εξελίσσεται από μέρα σε μέρα το πράγμα δηλαδή. Μαρία Τολπάνεν. Από τη Φιλανδική Βουλή. Όχι, ε, Ευρωβουλευτή από τη Φιλανδία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ολόκληρη ημέρα ε, συζητούσαμε για τους πρόσφυγες, ε, αλλά θα ήθελα να τονίσω ένα συγκεκριμένο πράγμα. Πρέπει να σκεφτούμε ποιοι είναι αυτοί οι πρόσφυγες. Έχουμε κρίση προσφύγων ή κρίση ετούντων άσυλο. Είναι διαφορετικά αυτά τα δύο. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να ξέρουμε ότι το βάρος του προπολογισμό είναι τεράστιο. Είναι οι πρόσφυγες που έρχονται στην Ευρώπη χωρίς εργασία και μπορεί να ζητήσουν επίδομα ανεργίας ας πούμε. Και αυτό αποτελεί ε, μεγάλο πρόβλημα. Ειδικά στα κράτη στα οποία υπάρχουν ε, πολλές, ε, πολλοί μηχανισμοί προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας. Είναι προβληματική η κατάσταση και κοστίζει. Αν θέλουμε όλα αυτά τα προβλήματα να τα λύσουμε ταυτόχρονα να Ένωση είναι δύσκολο. Δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε και γι' αυτό πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες. Τώρα, προς τα πού θέλουμε να το πάμε το ζήτημα. Στη Φιλανδία ε, πιστεύουμε ότι το κάθε πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίζεται ε, χωριστά. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Δεν μπορούμε να κρατάμε πολλά καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να θέσουμε προτεραιότητες. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των, των ετούντων άσυλο ή των προσφύγων. Θέλουμε να μιλήσουμε για ειρήνη. Τι θέλουμε. Αυτό είναι το α και το ω νομίζω η ειρήνη. Και η αλλαγή του κλίματος ε, θα φέρει και αυτή πολλές αλλαγές. Σκεφτείτε, με την άνοδο των υδάτων. Θα υπάρχουν περιοχές στην Ασία που θα πλημμυρίσουν και αυτό δεν πρέπει να μας ε, εκπλήσει. Ε, δεν πρέπει να μας εκπλήσει καθόλου, όπως δεν πρέπει να μας εκπλήσει και η κρίση των ετούντων ασύλων. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την αλλαγή του κλίματος, ας πούμε, να πω σύντομα. Στην Φιλανδία είχαμε τρία μέτρα χιόνι στο παρελθόν. Τα παιδιά έπρεπε να σκάψουν για να περπατήσουν και τώρα απλώς βρέχει το χειμώνα. Έτσι, σύντομα, πριν λίγα χρόνια ήταν αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις μεταφορές για την σοφροσύνη. Τώρα, επόμενη ομιλήτρια, Ιζαμπέλ Πυρές, από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Μπλόκο Ντεσκουάρντο. Εσκουερντά. Κέρδα. Διορθώνει. ζητώ συγγνώμη. Καλό απόγευμα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι με τη συζήτηση αυτή μπορέσαμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα για τον προϋπολογισμό και την επικουρικότητα. Υπάρχει ένα πλαίσιο προϋπολογισμών, αλλά υπάρχει και ένα πολιτικό πλαίσιο. Υπάρχουν θέματα τα οποία απαιτούν άμεση απάντηση και μια κοινή απάντηση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την κρίση του προϋπολογισμού και την χρηματοοικονομική κρίση, αλλά συγχρόνως και μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση και την κρίση του Σέγγεν και επίσης όλα αυτά τα ιδεολογικά προβλήματα που έχουν οδηγήσει στην τεράστια ανεργία των νέων στην Ευρώπη. Αυτό είναι φανερό ότι χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις και είναι φανερό ότι χρειάζονται περισσότερες συζητήσεις για τα θέματα αυτά αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε να δούμε ποιε είναι οι πολιτικέ προτεραιότητε που θέλουμε να δώσουμε στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή θα είναι ίσω μια από τι κέρδε συζητήσει για τι πολιτικέ ε, συζητήσει. Μέσα στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα λοιπόν να σταθώ στο θέμα τη ανεργία των νέων που είναι γνωστό ότι έφτασε πάρα πολλά, πολύ ψηλό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες όπως η Πορτογαλία έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο. Θα πρέπει λοιπόν η πρωτοβουλία για τους νέους να μπορέσει να αναστρέψει αυτή την τάση, να βοηθήσει τους νέους και να εμποδίσει τους νέους να βρισκόνται στην ανεργία ή σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Υπάρχουν όμως δύο βασικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σχετικά. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος αυτού για το 2016 γιατί δεν έχουμε ακόμα την σαφήνεια για το κατά πόσον θα μπορέσουμε να, δεν έχουμε και τρόπο να δούμε κατά πόσον έχει γίνει σωστά η βελτίωση της απασχόλησης των νέων και παραμένουν σε υψηλό επίπεδο η, τα επίπεδα Επίσης το δεύτερο ερώτημα που συνδέεται είναι τι είδους εργασίας θέλουν οι νέοι και αν είναι επαρκής μια εργασία η οποία είναι επισφαλής. Ένα τελευταίο σημείο το οποίο θέλω να θέξω να θέσω είναι σε σχέση με την κατάσταση των προσφύγων. Ενώπιον τη κατάσταση των προσφύγων, στο Πορτογαλικό Κοινοβούλιο συζητήσαμε ιδιαίτερα για τα ζητήματα αυτά και πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το αντικείμενο τη επόμενη συζήτηση, λέει ο πρόεδρο. Σα ζητώ συγγνώμη. Να σα πω το εξή πάρα πολύ εν συντομία ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουν όλοι. Υπάρχει η ανάγκη να εξασφαλιστεί μια ισορροπία και να ενθαρρύνουμε και πάλι την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να έχουμε χώρες οι οποίες υφίστανται όλο το βάρος της προσφυγικής ζωής, ενώ άλλες δεν κάνουν τίποτα. Θα πρέπει να βρούμε απαντήσεις σε αυτό και επίσης να δώσουμε μεγαλύτερη βοήθεια σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία που αντιμετωπίζουν ένα υπέρμετρο βάρος και επομένως δεν πρόκειται μονάχα για χρήματα, αλλά πρόκειται και για υποστήριξη σε επίπεδο αλληλεγγύης και υποστήριξη για να βελτιωθούν και τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων. Ευχαριστώ. Ο, Ραλφ Μπριγκ Χάους από την Bundestag και ο οποίος είναι στην ε, αντιπροσωπεία του ΕΛΚ, στη γερμανική αντιπροσωπεία του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο για το θέμα της χρηματοδότησης των προσφύγων. Ε, με εκπλήσει λίγο το γεγονός ότι αναφέρθηκε τόσες φορές ε, το παράδειγμα των προσφύγων που αφήνονται να υποφέρουν ε, και υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που ήρθαν στην Γερμανία και στην ε, Σουηδία. Αυτέ οι χώρε παίρνουν όλο το βάρο. Ε, και όλε οι άλλε χώρε απλά θέλουν να του στείλουν όσο πιο γρήγορα γίνεται σε αυτέ τι ε, χώρε. Το παράδειγμα του Καλέ. Δεν είναι η Γαλλία δυστυχώ κατά τη γνώμη μου μια χώρα που υποφέρει από του πρόσφυγες. Και πραγματικά εκπλησόμαστε. Ποιε είναι αυτέ οι χώρε που αναφέρουν τώρα ότι πρέπει να αλλάξουμε το σύμφωνο ε, το δημοσιονομικό για τους λόγω των προσφύγων. Ε, είναι η Γερμανία και η Σουηδία και ίσως και η Ιταλία που πλήττονται, αλλά όχι και άλλες χώρες κατά τη γνώμη μου. Η δική μας γενιά έχει υποχρέωση να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε μέσω χρεών για να υποφέρουν οι επόμενες γενναίες. Έχει δίκιο ο συνάδελφος από την Φιλανδία. Οι επόμενοι θα ασχολούνται με την καταστροφή του κλίματος και άλλες καταστροφές. Πρέπει λοιπόν επιγόντως να έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική για το χρέας και τελικά να λύσουμε το θέμα της κρίσης των προσφύγων. Τελευταία παρατήρηση. Θεωρώ ότι σίγουρα η Γερμανία έχει κάνει κάποια λάθη ως προς την ε, λήψη των ε, προσφύγων και των ετούντων άσυλο. Όμως το γεγονός είναι ότι ξεκίνησε να κινητοποιείται ο κόσμος και τώρα ε, είμαστε μόνο στην αρχή. Ε, δεν ξέρουμε αν θα είναι ένας φίλος πόλεμος ή οποιοδήποτε άλλος πόλεμος ή το κλίμα που θα έχουμε ως πρόβλημα στο μέλλον. Όμως από κοινού Ευρώπη πρέπει να έχουμε κοινή ευθύνη. Κάθε χώρα πρέπει να κάνει το δικό της μερίδιο και να βελτιστοποιήσουμε τις ε, λύσεις γιατί αλλιώς θα καταρρεύσει η Ευρώπη και οι άνθρωποι που έρχονται από την Αφρική και άλλες περιοχές ε, δεν θα έχουν καμία προοπτική. Δεν είναι θέμα μόνο χρημάτων. Στις 18 και 19 Φεβρουαρίου πρέπει να βρούμε μια κοινή απάντηση στο θέμα, γιατί αν δεν τη βρούμε δυστυχώς η Ευρώπη θα έχει τους επόμενους μήνες και τις εβδομάδες μάλλον ε, ένα πολύ ε, πήγον ζήτημα να αντιμετωπίσει. Σας ευχαριστώ για τη μαρτυρία. Έχετε το λόγο. θέλω να υπογραμμίσω το ανθρώπινο κόστος του τι συμβαίνει. Με τους νέους στην Ιρλανδία. Υπάρχουν ε, τεράστια ψυχολογικά προβλήματα. Οι νέοι είναι το επόμενο θέμα. Okay, sorry. Συγγνώμη. Bon, alors on va en rester euh, Αρκούν αυτά για τους πρόσφυγες, νομίζω. Φυσικά, οι συνθήκες υποδοχής στις ευρωπαϊκές χώρες, ε, η Γερμανία, Σουηδία, πρέπει να μιλήσουμε και για την Ιταλία και την Ελλάδα όμως, και για κάποιες άλλες χώρες. Αυτά συνιστούν τεράστιο πρόβλημα στην Ευρώπη, αλλά βεβαίως έχουμε και θέματα ε, και προβλήματα με την υποδοχή προσφύγων σε μη ευρωπαϊκές χώρες. Ε, Τουρκία, Λίβανο, Ιορδανία και η υποσαχάριος Αφρική. Ε, που υπάρχει και εδώ και θέμα ε, αναπτυξιακής πολιτικής. Είδαμε ότι η Σύνοδος της Βαλέτας Ε, Μα άφησε έτσι μια πικρή γεύση γιατί δεν θεωρούμε ότι έγινε ουσιαστική πρόοδος. Δεν, άλλαξε τίποτα. Παρακαλώ. ποιες είναι οι παρατηρήσει σας, κύριε Βαλιέ ε, και κυρία Ρεγκάνζο, ε, που θα κλείσουν και τη σύνοδο αυτή να πω στους Γερμανούς φίλους ότι εγώ δεν εκπροσωπώ κάποια κυβέρνηση. Μιλάω μόνο εξ ονόματος των περιφερειακών και τοπικών αρχών. Και έχω συνείδηση της προσπάθειας που έχει γίνει από τους ε, Γερμανούς δημάρχους, κυρίως του Μονάχου, αλλά θα μπορούσα να αναφέρω και το δήμαρχο της Βιέννης και πολλούς άλλους δημάρχους στην κεντρική Ευρώπη που έκαναν προσπάθεια για να υποδεχθούν τους πρόσφυγες. Θα ήθελα να πω επίσης ότι η αλληλεγγύη δεν είναι επιλογή στην Ευρώπη. Δεν είναι επιλογή είναι η ευρωπαϊκή δέσμευση, η οποία φέρει το πλαίσιο της αλληλεγγύης και αφορά όλες τις πολιτικές. Αλλά κυρίως για την υποδοχή των προσφύγων συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η βουλευτής από τη Φιλανδία, ότι αυτή η κρίση δηλαδή είναι ένας κρίκος μια συνολικής κρίσης που θα μας ακολουθεί τα επόμενα χρόνια. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή πολιτική ε, ασύλου και την δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, Ευρωπαϊκούς Οργανισμού για μια κοινή πολιτική ασύλου και υποδοχής προσφύγων. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, είναι απαραίτητο. 28 ε, χώρες σημαίνει 28 διαφορετικές αντιλήψεις ε, για την υποδοχή. Ε, φαντάζεστε τι πρόοδο έχουμε να σημειώσουμε. Ε, ως Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου ε, Δήμων και Κοινοτήτων της Ευρώπης είναι, το μήνυμά σας είναι ότι ένα τμήμα των διαστατικών ταμείων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπίσουμε τι, την υποδοχή των προσφύγων με σωστές συνθήκες. Γιατί αλλιώς δεν θα τα καταφέρουμε. Κοιτάξτε, δεν γίνονται θαύματα. Η Ευρώπη δεν γεννάει χρήμα. Με τα ταμεία που έχουμε και με τα κονδύλια που έχουμε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι προτεραιότητε. Και τι θέλετε να μου πείτε ότι η υποδοχή ας πούμε, των προσφύγων δεν είναι προτεραιότητα, είναι ε, ας κάνουμε λιγότερου ποδηλατόδρομου και λιγότερου αυτοκινητόδρομου τελικά. Αυτό σημαίνει ότι, έχουμε, ότι η υποδοχή των προσφύγων είναι προτεραιότητα. Λοιπόν, η κυρία Ρόι Γκραζό υποστηρίζω αυτή την τελευταία παρέμβαση. Ε, ένας μηχανισμός πιο άμεσης πρόσβασης ε, για την πρόσβαση των ταμείων από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, αυτό θα ήταν ένα καλό στοιχείο, θα ήταν πρόοδος. Και κάτι πιο συγκεκριμένο. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δια, διαπραγματευτούμε με τον ε, Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης για να αναπτύξουμε ένα δυναμικό υποδοχής 1.500 ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη. Πέρα από όλα όσα έχουν γίνει για να φτάσουμε στα νούμερα που διαπραγματευτήκαμε στο 28 στις 29 συγγνώμη, Οκτωβρίου. Ε, και αν υπήρχε μια σιγουριά ότι θα υπήρχε άμεση χρηματοδότηση, χωρίς να περάσουμε από 200 ας πούμε παρατρεχάμενους, ε, αυτό θα ήταν πολύ καλό και θα μπορούσαμε να πάμε πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο ευέλικτα μπροστά. Επομένω, θέλω και εγώ με αυτή την παρέμβαση να υποστηρίξω τον, τον πρώτο τελευταίο μιλητή. Περνάμε στο τελευταίο κομμάτι οικονομικέ ανάγκε για να ξεπεράσουμε την οικονομική και κοινωνική κρίση. Ε, παράδειγμα, ε, η εγγύηση των νέων. Έξι ώρα κλείνουμε. Έχουμε 45 λεπτά και όχι μία ώρα λοιπόν. Άρα, Κυρία Ιντσέρτη, παρόλα αυτά, εσεί έχετε, έχετε συγκεκριμένο χρόνο. Είσαστε μέλο τη Επιτροπή Απασχόληση ε, τη Ιταλική Βουλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω πολύ γρήγορα ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο έτσι το υπενηχθήκαμε. Θα ήθελα να θέσω έτσι στο κέντρο μιας ευρωπαϊκής δράσης που χρειάζεται. Εσείς μιλήσατε για ένα προγράμματα το οποίο έδωσε καρπούς σε απάντηση όλων αυτών που ζητούσαν να δουν τι δυναμικό έχουν οι, ε, τα ευρωπαϊκά ταμεία ε, και πόσο μπορούν να προωθήσουν ας πούμε, μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα. Ε, το παράδειγμα είναι η εγγύηση για τους νέους. Ειδικά ε, για τις περιοχές εκείνες όπως την Ιταλία που έχουμε τεράστια ενεργεία, πάνω από 25%. Μιλάμε για παιδιά 15 ε, έως 24 με 25 χρόνων. Ε, και μιλάμε για την εκπαίδευση, απασχόληση και κατάρτιση. Έτσι. Τώρα που θα γίνει η αναθεώρηση του προπολογισμού, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό είναι ένα μέτρο που κατά τη γνώμη μας πρέπει να υποστηριχθεί και να το χρηματοδοτήσουμε και στη συνέχεια. Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Επιτροπής Προπολογισμού που είναι την ευκαιρία να παρέμβω εδώ για να μιλήσω για την ανάγκη να παρατείνουμε ε, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία που ονομάζεται εγγύηση για τους νέους. Και είναι πολύ σημαντικό το ενδιαφέρον που δείχνουμε για αυτό το μέτρο που θεωρώ πάρα πολύ καινοτόμο και που ξεκίνησε το 2013 πριν τρία χρόνια. Και θα κάνω και κάποια έτσι γενικά σχόλια, κάποιους προβληματισμούς που νομίζω είναι χρήσιμοι. Και θα δώσω και κάποια στοιχεία για να σας δείξω την εμβέλεια αυτής της προσπάθειας, αυτής της πρωτοβουλίας. Να προσθέσω ότι αυτό δεν αφορά μόνο κάποιες χώρες, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και όχι τη Γαλλία. Θέλω να υπενθυμίσω ότι οι μακροοικονομικές προβλέψεις ε, του χειμώνα που εκδόθηκαν πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή δείχνουν ξεκάθαρα ότι φτάσαμε στην τέταρτη χρονιά ανάκαμψης ξεπεράσαμε την πιο οξία φάση της κρίσης, αλλά παρόλα αυτά δεν νομίζω ότι ακόμα έχουμε σημάδια μιας ανάπτυξης αρκετά ισχυρής, ούτως ώστε να υπάρχει σοβαρή μείωση της ανεργίας, κυρίως των νέων. Οι επενδύσεις ανακτούν τη δύναμή τους βέβαια, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτό που θα θέλαμε να είναι. Όπως ε, είπαμε και σήμερα το πρωί, είμαστε στο 1,9% ε, φέτος ε, των συνολικών, δηλαδή επενδύσεις, στο, και, πέρυσι, και πέρυσι το ίδιο, 1,9%. Δηλαδή, ε, συγγνώμη, το 1,9% είναι ε, ποσοστό ρυθμός ανάπτυξης πολύ χαμηλός. Έχουμε μια πολύ έτσι μέτρια βελτίωση της κατάστασης ε, που θα έπρεπε στην ε, Ευρωζώνη να μειώσει την ε, ανεργία και να τη φτάσει γύρω στα 10%. Στην Ευρωζώνη πάντα. Και για την ανεργία των νέων, παρότι έχουμε μια αντιστροφή της πορείας, παρόλα αυτά ακόμα είναι πολύ ψηλή Έχουμε δεδομένα του Δεκεμβρίου του 2015. Έχουμε ποσοστά αργίας των νέων 20-21% στην Ευρωπαϊκή Μείωση. Σημαντική μείωση σε σχέση με πέρυσι, παρόλα αυτά δεν αρκεί σε σχέση με αυτά που είχαμε στο παρελθόν για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να δημιουργηθεί αυτό που λέμε η χαμένη γενιά, η οποία θα παγιδευτεί μέσα σε αυτή την ανεργία. Πολλοί από τους νέους ε, έχουν φύγει από τη σχολική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να σας πω πολύ γρήγορα ποια είναι τα βασικά αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας στην Ιταλία, ούτως ώστε να σκεφτούμε μαζί τα μέτρα που υιοθετήθηκαν και τις επιπτώσεις που αποδίδουν, που δίνουν. Το πρώτο θετικό στοιχείο αυτή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας, σε ό,τι αφορά την ε, απασχόληση των νέων, είναι η δυνατότητα να δημιουργηθεί διάλογος, μια ανταλλαγή πληροφοριών για τις ε, βέλτιστες πρακτικές που έχουμε αναπτύξει σε εθνικό επίπεδο. Ούτως ώστε να μάθουμε μένα από τους δε. Ξέρετε ότι η Ιταλία είναι η δεύτερη χώρα που υποφελείται από τους πόρους ε, της εγγύησης ε, για την νεολαία. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία. 560 ε, εκατομμύρια ευρώ. Σημαντικό ποσό. Φυσικά, αν ε, αντιπαραθέσουμε την ε, ανεργία των νέων στην Ιταλία, παρότι μειώθηκε, μειώθηκε κατά 1% την τελευταία χρονιά, το Δεκέμβριο όμως του 2015 βρισκόμαστε ακόμα στο 37,9%. Οι πόροι που είναι στη διάθεσή μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπήκαν σε ένα εθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα που το λέμε PON, ε, αρμόδιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο έχει ε, κινητοποιήσει συνολικά, έτσι, ε, πέρα από τα 567 εκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ε, και Ιταλικά, την εθνική δηλαδή συγχρηματοδότηση και φτάσαμε στο 1,5 δις στην Ιταλία. Τώρα κάποια στοιχεία για το ποιο συμμετείχε σε αυτό το πρόγραμμα. Ένα 1.720.000 ε, από 15 έως 29 ετών. Έχουμε επεκτείνει την, την ψαλίδα αυτή λόγω του ότι έχουμε ε, πολλούς μακροχρόνια άνεργους, νέους άνεργους ε, που δεν ούτε πάνε σχολείο, ούτε πάνε στο πανεπιστήμιο, ούτε ε, εργάζονται. Και έδειξαν ενδιαφέρον να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. είναι πολύ πρόσφατα στοιχεία μας τα δίνει το Υπουργείο, ε, το οποίο επικαιροποιεί το site του ε, μηνιαίως και δείχνει, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι ένα εκατομμύριο νέοι περίπου ε, εντάχθηκαν και συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα. Πάνω από το 50% λοιπόν των ενδιαφερόμενων νέων 15 με 29 ετών γράφτηκαν και έδειξαν ενδιαφέρον. Ε, ο αριθμός των νέων οι οποίοι πραγματικά βρήκαν δουλειά είναι 600.000. Ε, τα στοιχεία τα έχετε στη διάθεσή σας. Αυτό σημαίνει ότι σε εμά ο αριθμός των καταγεγραμμένων νέων ε, συνεχίζει να αυξάνεται 10.000 ε, το μήνα όχι 10.000 τη βδομάδα μιλήτρια. Ε, Καινούργοι νέοι εγγράφονται στο πρόγραμμα αυτό. Αυξάνονται λοιπόν οι εγγραφές και αυξάνεται η συμμετοχή με ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό. Τον Ιανουάριο του 2015 είχαμε ποσοστά ε, που είχαμε 5% ε, αύξηση των ε, εγγραφών. Τώρα έχουμε 6% αύξηση των εγγραφών. Και από όλους όσους καταγράφονται, ε, λαμβάνουμε, δεχόμαστε μάλλον στο πρόγραμμα το 70% των νέων. Από τη στιγμή που γράφονται οι νέοι, μέχρι τη στιγμή που τα εργασία ευρέσεως, ε, τα ευρέσεως εργασίας ε, αναλαμβάνουν αυτούς τους νέους, ε, μειώνεται όλο και περισσότερο. Δηλαδή πολύ πιο γρήγορα ε, ενσωματώνουμε αυτούς τους νέους. και πολύ πιο γρήγορα ε, δίδεται απάντηση σε αυτούς τους νέους. Οικονομικός πώς υιοθετήθηκαν μέτρα και με βάση τα δεδομένα του Υπουργείου Εργασίας αφορούν, έχουμε ξοδέψει πάνω από τα 80% των ε, ποσών που ήταν στη διάθεσή μας. Έχουμε απορροφήσει δηλαδή. Αυτά τα νούμερα δείχνουν ότι αυτή η πρωτοβουλία προοδευτικά υλοποιεί τους στόχους, παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρότατε διαφορές ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες. Το θέμα βεβαίως της ε, εκπαίδευσης κατάρτισης ε, συνδέεται και με το πώς οι περιφέρειες ε, αναπτύσσουν και ερμηνεύουν αυτή την έννοια και η εγγύηση των νέων αποτέλεσε ένα στοιχείο, μια αφορμή για να ξαναδούμε τις πολιτικές μας και να προωθήσουμε τις ενεργητικές πολιτικές, γιατί πάντα ε, ήμασταν κολλημένοι στις παθητικές πολιτικές. Αυτός ο μηχανισμός ε, των νέων ε, έδωσε το πράσινο φως για να εργαστούμε και σε άλλα, πάνω σε άλλα μέτρα, ε, πάνω σε ενεργές πολιτικές. Έχουμε μια τεράστια διαδικασία μεταρρυθμίσεων στην Ιταλία, ε, μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, Jobs Act, ενεργές πολιτικές και χάρη στην εγγύηση των νέων, αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ευρέσεως εργασίας, ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια των υπηρεσιών προσφέροντας σε διάφορες περιφέρειες, μια νέα ε, οργάνωση, ένα οργανισμό σε εθνικό επίπεδο. Ε, αυτό λοιπόν το Youth Guarantee μας έδειξε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο, τουλάχιστον αυτό ήταν η δική μας εμπειρία, αλλά νομίζω ότι αυτό ισχύει και για τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες. Και αυτό είναι το πρώτο θετικό στοιχείο. Πρέπει να κλείσω την παρέμβασή μου. Πολύ γρήγορα. Σα παρακαλώ λίγο λίγο, ε, σιγά σιγά φτάστε στο συμπέρασμα στο οποίο θα την καταλήξετε. Έχω πάρα πολλά να πω ακόμα, αλλά τι να κάνω. Καλά είναι και αυτά που είπα. Όλα αυτά τα στοιχεία που σας δίνουν, σας δείχνουν ότι η διαδικασία αυτή είναι εξελίξη, πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Είναι θετικά όμως τα πρώτα στοιχεία είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η πρώτη αξιολόγηση είναι θετική. Ακόμα και συμβολικός πώς. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με περιορισμένους πόρους, το οποίο όμως δίνει απτά αποτελέσματα και πραγματικά δείχνει στους πολίτες τι είναι στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να προωθήσει τη μεγαλύτερη, μια μεγαλύτερη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Σε αυτή τη φάση που μόλις βγήκαμε από την οικονομική κρίση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχετε φυσικά την ευκαιρία να απαντήσετε στα διαφορά ερωτήματα. Κύριος που είχα διακόψει σας ξαναδίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πολλά να πω και για τους πρόσφυγες, αλλά θα μιλήσω για το θέμα των νέων. Η ανεργία των νέων στην ε, Ιρλανδία είναι πραγματικά τρομερή. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας των νέων μέσα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η μόνη ελλακτική λύση που έχουν αυτή τη στιγμή και φυσικά αντιμετωπίζουν και πολλά προβλήματα ψυχικής υγείας οι νέοι οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Τους είπανε είτε να πηδήξουν στο ποτάμι και να πνιγούν ή να πάρουν ένα αεροπλάνο και να φύγουν. Έχουμε χιλιάδε ανθρώπων, οι οποίοι νέων ανθρώπων που φεύγουν από την Ιρλανδία και μεταναστεύουν για να βρουν καλύτερη τύχη και είναι σκάνδαλο ότι η εγγύηση για του νέου δεν έχει λειτουργήσει, δεν υπάρχει καμία δέσμευση για να δοθεί αυτή η υποστήριξη. Έχουμε και συστήματα για παροχή απασχόληση που δίνουν ψίχουλα μόναχα. Κοστίζει να πάρεις μια τέτοια δουλειά και όχι και δεν βγάζει λεφτά. Έχουμε προβλήματα με απομόνωση ορισμένων περιοχών της υπαίθρου και σίγουρα αυτή η ανάκαμψη, αν υπάρχει μια τέτοια ανάκαμψη, σίγουρα δεν την έχουν καταλάβει οι νέοι στην Ιρλανδία. Και δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτοί οι οποίοι θα κληρονομήσουν την Ευρώπη τους έχουμε βάλει στο περιθώριο με τέτοια ευκολία. Λες και αυτοί έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει περισσότερη πίεση στα εθνικά κοινοβούλια και ιδίως όταν πρόκειται για την αξιολόγηση, να μην θεωρείται ένα δευτερεύον θέμα και να μην ξαναγυρίσει ποτέ. Χρειαζόμαστε να έχουμε τις σωστές κοινωνικές δομές, χρειάζεται να έχουμε τους κατάλληλους πόρους, την κατάλληλη κατάρτιση για να εξασφαλίσουμε ότι οι νέοι μας θα έχουν κάποιο μέλλον, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουν στη Ιρλανδία κανένα τέτοιο μέλλον. Ο Βλαδίμηρος Μάνκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα πολλές θετικές ε, ιδέες για αυτό το θέμα. Στην Σλοβακία για παράδειγμα χρηματοδοτήθηκε το πρόγραμμα αυτό ένα συγκεκριμένο project και στο τέλος ε, του project το 86% των ανθρώπων που συμμετείχαν σε αυτό είχαν δουλειά. Ήταν επιτυχημένο. Όμως για τον προϋπολογισμό του 2016 κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων το Συμβούλιο είπε ότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε δεσμεύσεις για αυτό το έτος γιατί αυτό το ε, project δεν έχει αξιολογηθεί. Ευτυχώς στυλώσαμε τα πόδια και είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει τώρα η αξιολόγηση, το 2015 δηλαδή. Δυστυχώς ακόμα δεν έχει γίνει η αξιολόγηση αυτή. Αλλά τι θέλω να πω. Ε, πώς μπορεί το Συμβούλιο να ε, παίρνει τέτοιες αποφάσεις και να λέει ότι αυτό το project είναι μια επιτυχία που δεν έχει ακόμα χαρακτηριστεί επιτυχημένος επιτυχία και να σταματάει ένα τέτοιο project που τελικά είναι τόσο επιτυχημένο και δίνει ανάπτυξη και απασχόληση. Πρέπει να υπάρχει μια αλληλεγγύη ανάμεσα στο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια για να δείξουμε στο Συμβούλιο ότι η δική του θέση δεν είναι αυτή η μόνη που μετράει στη διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Ιζαμπέλ Πυρές που πριν ανέφερε το θέμα της απασχόλησης των νέων. Θα ήθελε να επανέλθει για να ξαναμιλήσει για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να επανέλθω στην προβληματική που θέλησα να ξεκινήσω σε λάθος σε χρονική στιγμή για την ανεργία των νέων θα ήθελα να αναφερθώ στα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε αυτή η πρωτοβουλία για τους νέους. Ποιο ήταν το απτό αποτέλεσμα του προγράμματος αυτού. Ακούσαμε και το παράδειγμα της Ιταλίας προηγουμένως και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε και άλλες εμπειρίες για το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών. Εξακολουθούν παρά την εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας να είναι άνεργοι πολλοί νέοι να έχουν θέσει εργασία σε απόλυτη επισφάλεια. Το θέμα λοιπόν της ε, γνώσης του τι έγινε στα διάφορα κράτη-μέλη είναι πολύ ενδιαφέρον για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Και επίση μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα το είδο ε, θέσεων εργασία που έχει δημιουργηθεί με αυτήν την πρωτοβουλία για την εγγύηση των νέων. Γιατί σε πολλέ περιπτώσει, σε πολλέ χώρε, απλώ δημιουργήθηκαν επισφαλεί θέσει εργασία και επομένως δεν δίνουν κανένα μέλλον, δεν δίνουν καμία <clears throat> ελπίδα στους νέους όπως είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια. Σε συγκεκριμένες λοιπόν περιπτώσεις οι νέοι περνάνε από μία μαθητεία σε μία άλλη μαθητεία και δεν βρίσκουν ποτέ θέση εργασίας με το θέμα αυτό. Αυτό επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν το μέλλον και ίσως θα, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αναθεωρηθεί όλη αυτή η πρωτοβουλία γιατί δεν μπορεί με τον τρόπο αυτό να επιλύσει διαφθορτικά προβλήματα ανεργίας. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος είναι να υπάρχουν πραγματικές παρεμβάσεις οι οποίες θα αντιμετωπίσουν τα διαφορετικά θέματα. Είναι λοιπόν το ερώτημα αν στον προϋπολογισμό θα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να θεωρηθεί η απασχόληση των νέων μία από τις μεγάλες προτεραιότητες και φυσικά μια απασχόληση με δικαιώματα, με αξιοπρέπεια, γιατί και αυτό το θέμα δεν μπορούμε να το αφήσουμε απ' έξω μέσα στη συζήτηση για μια πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Δεν έχω άλλους οι οποίοι να θέλουν να λάβουν το λόγο. Κυρία Ιντσέρτη, Ίσως μπορείτε να απαντήσετε, αλλά εφόσον έχουμε και λίγο χρόνο, θα ήθελα να ξεφύγω λίγα από λόγο, από το ρόλο μου ως Προέδρου και να παρέμβω ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι γεγονός ότι η ανεργία των νέων έχει υποσκάψει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ένας στους τέσσερις νέους είναι άνεργος σε ορισμένε χώρες, ο ένας στους δύο. Εκτός τις λίγες χώρες που έχουν βαθιά ριζωμένες παραδόσεις στον οικονομικό ιστό, στην τοπική κουλτούρα, την μαθητεία. Αυτό βλέπουμε στη Γερμανία, αυτό βλέπουμε στις κάτω χώρες, αυτό βλέπουμε στην, στην Αυστρία. Και κάποιοι από εμά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε υπερψηφίσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να αυξήσουμε, να ενθαρρύνουμε την ε, κινητικότητα των νέων. Γιατί η εμπειρία μας είναι ότι αυτοί οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει το σύστημα Εράσμους, και έχουν ε, περάσει και ένα χρόνο ή παραπάνω έξω από τη χώρα τους ε, είναι καλύτερα οχυρωμένοι έναντι του κινδύνου της αδρίας. Θα πρέπει λοιπόν να επιτρέψουμε σε αυτούς που βρίσκονται σε μαθητεία να μπορούν να περάσουν ένα χρόνο εκτός από την χώρα προέλευσής τους και να ενθαρρύνουμε την κινητικότητα των των. Είναι δύσκολο λοιπόν να μπορέσουμε μέσα στο πλαίσιο των 28 ευρωπαϊκών χωρών να εναρμονίσουμε τους κανόνες για τη μαθητεία. Σε ορισμένε χώρες δεν υπάρχει κανένας κανονισμός για αυτές τις μαθητείες. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε σε τέτοια συγκεκριμένα μέτρα και να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει σύγκληση των ρυθμίσεων για την μαθητεία. Δεν μπορούμε να έχουμε μια εσωτερική αγορά με 28 διαφορετικές ρυθμίσεις. Και αυτό ισχύει φυσικά και για άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις όπως το δημοσιονομικό τομέα στον φορολογικό. Θα ήθελα λοιπόν να υπενθυμίσω στους εθνικούς ε, βουλευτές ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το κάνουμε και έχουμε ενώπιον μας ένα πείραμα. Θα ζητήσει η Κομισιόν σε κέντρα ε, κατάρτισης για να υπάρξει μια διαδικασία υποβολής προτάσεων από τους νέους που μπορούν να προτείνουν τουλάχιστον δύο κέντρα σε άλλες χώρες αν γνωρίζουν καλά τη χώρα της προέλε, της, της, την χώρα υποδοχής να μπορέσουν να προχωρήσουν σε μια θεωρητική κατάρτιση η οποία θα βοηθήσει τους νέους αυτούς και επίσης να συνδεθούν με ένα δίκτυο επιχείρησεων που μπορούν να υποδεχτούν αυτούς τους νέους ως ως μαθητιώντες. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τα εμπόδια και τις τροχοπέδες για την κατάρτιση και την κινητικότητα των μαθητευομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζουμε ότι αυτή είναι μια δυνητική απάντηση που θα επιτρέψει στους νέους να πλησιάσουν τον απόμακρο χώρο της εργασίας. Αυτή ήταν η τελευταία μου λοιπόν παρέμβαση και σας δίνω τον λόγο. Sì, e, Φυσικά, έκανα απλώς ποσοτικές αξιολογήσεις εγώ μόνο. Και αυτό είναι μια, μια μικρή ψηφίδα ε, από το γενικότερο μοσαϊκό του πώς θα αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων. Και κυρίως τι, ποια είναι τα διαφορετικά μέτρα ε, βιομηχανικής πολιτικής, επενδύσεων, που είναι τα πρώτα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Απλώς θα τονίσω ότι αυτό το μέτρο είναι ένα από τα λίγα, φυσικά στο συζητήσουμε, και προφανώς αυτό επέσυρε άλλα μέτρα στο χώρο. Παραδείγματο χάρη τώρα έχουμε ε, υποτροφίες ε, για την ε, κατάρτιση. Οι υποτροφίες είναι ένα από τα στοιχεία, το, το βασικό στοιχείο που θα επιτρέψει στον νέο να μπει στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν όμως και άλλα μέτρα, όπως παραδείγματο χάρη της κατάρτισης. Εδώ μιλάμε, μην ξεχνάτε, για κάποια μέτρα τα οποία αφορούν άτομα τα οποία δεν πάνε πια σχολείο και δεν έχουν ε, καν επαφή με την αγορά εργασία. Δηλαδή, η μαθητεία λοιπόν είναι ε, ας πούμε ένα σκαλοπάτι για να βοηθήσει τον νέο να μπει στην αγορά εργασία. Επίσης, ε, αυτές οι συμβάσεις ε, μαθητείας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Εμείς την έχουμε αναπτύξει αυτή την έννοια, τη χρησιμοποίησαμε πάρα πολύ χάρη σε αυτό το σχήμα της Ευρώπης εγγύηση ε, για την νεολαία. Αλλά επίσης μέτρα για την αυτοαπασχόληση. Πολύ σημαντικό. Από μόνο, από του το μέτρο αυτό δεν αρκεί φυσικά. Θα πρέπει να το συνδυάσουμε με πολλά άλλα μέτρα. Και επίσης αυτό που θέλω να τονίσω είναι παρά τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, πρέπει να δούμε πού πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις. Παρόλα αυτά θα ήταν λάθος να μην, καταρτήσουμε, να μην καταστήσουμε αυτό το μέτρο διαρθωτικό. Θα ήταν λάθος η κοινότητα, η Ένωση δηλαδή, τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια να μην συνεχίσει αυτό το μέτρο. Γιατί θα χάναμε όλους αυτούς τους πόρους, που δεν είναι και πάρα πολλοί, που κρατήσαμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, θα χάσουμε δηλαδή αυτού τους πόρους που δώσαμε αρχικά. Φυσικά το θέμα της αγοράς εργασίας, το θέμα της βιομηχανικής πολιτικής, το θέμα της ε, επενδυτικής πολιτικής, όλα αυτά είναι πολύ πιο θέμα, ευραία θέματα. Ζητώ συγγνώμη, εγώ μόνο άγγιξα την ε, το θέμα που αφορά την συνέχιση αυτού του μέτρου. Ε, το, το μέτρο δηλαδή που αφορά την εγγύηση για τους νέους. Να συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Φτάνουμε στα συμπεράσματα. Μετά από ανταλλαγές απόψεων που ήταν ιδιαίτερα εμπλουτιστικές και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου. Η κυρία Τομά έχει εμπλακεί στην προετοιμασία της μεταρρύθμισης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και ελπίζω ότι μπόρεσε να βρει και κάποιες πρόσθετες πληροφορίες για να βελτιώσει το έργο της και να προετοιμάσει την έκθεση που θα διαμορφώσει μαζί με τον κύριο Όλμπριχτ και που θα αποτελέσει αντικείμενο ψηφοφορίας, εξέταση και ψηφοφορίας από την Επιτροπή Προεπολογισμών τη, κατά τη διάρκεια της ε, άνοιξης. Θα είναι η άνοιξη του προϋπολογισμού, προϋπολογιστική άνοιξη. Βρισκόμαστε στο τέλος ενός κύκλου. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Άλλο. Εκτός αν θέλουμε να δείξουμε την ανικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους Ευρωπαίους πολίτες. Θα υπάρξουν πολλοί κίνδυνοι αν παραμείνουμε σε αυτή την εικόνα αδυναμίας και ανικανότητας. Κύριε Τωμά, μήπως θέλετε να μας δώσετε ορισμένα συμπεράσματα, καταληκτικά. Με μεγάλη ταπεινοφροσύνη θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τον κύριο Βαλιέ και την κυρία Ζώζα και την κυρία Ινσέτη για τη συμμετοχή τους και την συμβολή τους. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες που μας έφεραν, όπως είπατε, από όλους τους ε, παρόντες και θα τις εξετάσουμε βέβαια μεταξύ των προτάσεων αυτών Υπάρχουν κάποιες οι οποίες θα απαιτήσουν μεταρρύθμιση των συνθηκών. Ενδεχομένως μπορούμε να τις αναφέρουμε. Α, ο κύριος Κάμερον ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει, λέω ο πρόεδρος. Ναι, αυτή είναι καλή ιδέα. Υπάρχουν κάποιες ιδέες οι οποίες μπορούν να έχουν χαρακτήρα απότερων προοπτικών, αλλά και υπάρχουν και ιδέες οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και σε επίπεδο όχι εθνικό αλλά εδαφικό, να μπορέσουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να έχουν άμεση πρόσβαση στον προϋπολογισμό και στη συνέχεια υπάρχουν πολλές συζητήσεις οι οποίες γίνονται στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Τα έχουμε συζητήσει ήδη τα θέματα αυτά. Δυστυχώς δεν είναι πολύ ο κύριος Όλμπριχτ εδώ, αλλά νομίζω πρέπει να σκεφτούμε και τους κανόνες του παιχνιδιού. Όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους των Ταμείων Συνοχής πρέπει να σας πω ότι οι κανόνες του, των πολιετών, του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 είναι ήδη σαφής. Δεν μπορούμε να πειράξουμε τα εθνικά ποσά μέσα στα ταμεία συνοχής που έχουν ήδη καθοριστεί. Ναι, θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι σε αυτή την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου γιατί είδαμε ότι ο, το πλαίσιο 2014-2020 δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες, αλλά υπάρχουν και κανόνες στους οποίους πρέπει να τους σεβαστούμε. Για αυτούς τους λόγους δεν μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μαγικό ραβδάκι για να λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας των νέων. υπήρξε η έλβηση του Κοινοβουλίου που ζήτησε να υπάρξει ένα ειδικό ταμείο το οποίο θα έπρεπε να δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Και δεν μπορούμε παρά να λυπηθούμε ότι μετά από δύο χρόνια που έχει τέθει σε εφαρμογή αυτή η διαδικασία ουσιαστικά έχει ανασταλεί αυτή η διαδικασία. Αυτό δεν δείχνει ιδιαίτερη σοβαρότητα για να το πω ούτως. Έχουμε πολλά πράγματα λοιπόν να συζητήσουμε. Εν πάση περιπτώσει τα έχω σημειώσει όλα αυτά που είπατε και μην διστάσετε να συμβάλλετε και γραπτά εάν θέλετε να μου φέρετε κάποιες ιδέες για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και μην λησμονήσατε, το λέω και για την συνάδελφο από την Φιλανδία είναι πάρα πολύ σημαντικό να καθορίσουμε σαφώς τις προτεραιότητές μας γιατί οι γραμμές του προπολογισμού που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες περικοπές το 2014-2020 είναι ακριβώς αυτές όπου χρειάζεται να επανέλθουμε στον προπολογισμό. Λοιπόν, κανένα εθνικό προπολογισμό έχει μία μοναχα πολιτική προτεραιότητα. και αν ε, κόψουμε τελείως μια δημόσια παρέμβαση στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε πώς θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη κρίση. Πρέπει λοιπόν από τη μια πλευρά να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που είναι κατεπίγοντα, αλλά από την άλλη μεριά να εξετάσουμε και τη διάθεση του προπολογισμού. Αυτό θα κάνουμε κιόλα. Κλείνουμε λοιπόν αυτήν εδώ την Διακοινοβουλευτική ε, Επιτροπή. Και η προσωπική μου ευχή είναι να μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τις συναντήσεις μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το δικό μας πρόβλημα ως Ευρωβουλευτές είναι ότι η Ευρώπη δυσκολεύεται να μιλήσει στους Ευρωπαίους. Και αν θέλουμε να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους τι ακριβώς είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, φοβάμαι ότι θα είναι δύσκολο. Βέβαια, η δημοκρατική απέτηση είναι να μπορούμε να θεσπίζουμε και να ψηφίζουμε έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που να είναι κατανοητός και εύκολος ε, για, τους, ε, για τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα έχουμε περιθώριο βελτίωσης ο προϋπολογισμός ως έκφραση μιας πολιτικής βούλησης και ενός οράματος ε, είναι εκεί ε, για αυτό το λόγο και μόνο και δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τα πάντα μέσα από τον προϋπολογισμό γιατί υπάρχουν θεσμικά προβλήματα και προβλήματα διακυβέρνησης. Άρα η Ευρώπη έχει πολύ σημαντικές πρόοδους να κάνει. Αυτό που θέλουμε να καταδείξουμε είναι ότι τα κονδύλια που χρησιμοποιούμε ε, μέσα στο προπολογισμό έχουν πραγματική χρησιμότητα. Ζητάμε από τα κράτη-μέλη να, να δώσουν μια εισφορά για να την πάρουν πίσω ε, τελικά μέσα από ένα αριθμιστικό πλαίσιο που είναι στενό σαν κορσές και δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς ε, πώς θα γίνει αυτό. Δεν μπορούν να καταλάβουν την πολυπλοκότητα, τη γραφειοκρατία και την αυθαιρεσία. Αυτό είναι το τέλος ενός κύκλου, μιας εποχής. Εμείς ως Ευρωβουλευτές που ασχολούμαστε με τον ε, προϋπολογισμό είμαστε ημιπληγικοί. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε πλήρως τα καθήκοντά μας. Εδώ δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα έσοδα, γιατί και τα κράτη-μέλη είναι και αυτά ε, περιορισμένα από τα 7 έτη και υπάρχει και μία καχυποψία, μία ιστερία για τις δαπάνες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνο και πρέπει ε, τώρα με την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου να αρθρώσει το λόγο του. Δυστυχώς όμως ε, δεν έχουμε κερδίσει το στοίχημα αυτό. Είναι οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων που αποφασίζουν. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή δημόσια γνώμη. Ελπίζουμε όμως ότι κάποια μέρα θα μπορούμε να απευθυνθούμε στους Ευρωπαίους για να μπορέσουν να δουν ποια είναι τα πράγματα που διακυβεύονται. Υπάρχει δυνατότητα αυτή της διαπραγμάτευσης, αλλά αυτός ο κορσές στην ουσία δεν μας αφήνει να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις κρίσης. Και γιατί δεν μπορούμε... Και όταν δεν μπορούμε μάλλον, ε, στην ουσία δίνουμε την εικόνα της ανικανότητας που τελικά τροφοδοτεί τον ε, λαϊκισμό και την ευρωφοβία. Άρα ήρθε η στιγμή να δείξουμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με την οποία είμαστε αντιμέτωποι, να θέσουμε προτεραιότητες και να κάνουμε και τους ε, διακανονισμούς ε, που χρειάζονται. Και αυτό είναι δείγμα πολιτικής επιδεξιότητας. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την συμμετοχή σας. Ο προϋπολογισμός είναι η εικόνα της πραγματικότητας. Στην πολιτική η πραγματικότητα συχνά είναι στην αντιπολίτευση. Ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλή τύχη.